Buenas tardes a todos y todas. Καλησπέρα σε όλους και όλες σας. Και στα γαλλικά και στα ισπανικά. Και στα αγγλικά. Dear colleagues, ladies and gentlemen. συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ για να αρχίσουμε. Καταρχάς θα ήθελα να σας καλωσορίσω στην κοινή ε, αυτή ακρόαση με τις δύο επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΑΦΚΟ. Έχουμε επίσης παρόντα μέλη από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, Γιούρι, ως συνδεδεμένη επιτροπή συμμετέχει. Επίσης, μέλη από την Επιτροπή Πολιτισμού και από την Επιτροπή Αναφορών έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν στην παρούσα ακρόαση. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε θερμά την υποψήφια αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία ε, Βέρα ε, Γιώροβα. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Ε, name of το χαρτοφυλάκιο σας, το υποψήφιο, έχει τον τίτλο «Αξίες και διαφάνεια». Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού μας, όπου προβλέπονται κατευθυντήριε γραμμές για την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Κοινοβούλιο πρώτα καλείται να αξιολογήσει την υποψήφια αντιπρόεδρο, τη γενική της επάρκεια, την ευρωπαϊκή τη προσήλωση, την προσωπική της ανεξαρτησία, καθώς επίσης και να εκτιμήσει ε, την γνώση της για τα θέματά της και τις ικανότητές της στην επικοινωνία. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, αφότου εξέτασε τη δήλωση οικονομικών συμφερόντων της υποψήφιας αντιπροέδρου, δεν προέβαλε αντιρρήσεις για τη διεξαγωγή αυτής της ακρόασης και γνωρίζουμε όλοι ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η συζήτηση θα γίνει ως εξής, ως ήθιστε. Η υποψήφια αντιπρόεδρος θα πάρει το λόγο για να κάνει μια εισαγωγή, λιγότερο από ένα τέταρτο της ώρας. Στη συνέχεια θα έχουμε το πολύ 25 ερωτήσεις από τους βουλευτές. Θα αρχίσουμε με τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων, οι εκπροσώπους, και μετά τα υπόλοιπα με μέλη που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο των ομιλητών για να κάνουν την ερώτησή τους. Μέχρι 25 συνολικά ερωτήσεις θα τεθούν. Με την ίδια δομή πάντα. Ένα λεπτό για την πρώτη ερώτηση Δύο λεπτά για την πρώτη απάντηση. Στη συνέχεια, ένα λεπτό συμπληρωματική ερώτηση, σχόλια. Και ένα λεπτό για την απάντηση. Το πολύ 25 ερωτήσεις. Και στο τέλος θα κλείσει η κυρία Γιούροβα. Θα αρχίσουν εκπρόσωποι, όπως είπαμε, των πολιτικών ομάδων, συντονιστές ή εκείνοι που εκπροσωπούν ε, τις ε, ομάδες τους. Σε 23 επίσημες γλώσσες θα έχουμε διερμηνία και παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι στην παρούσα ακρόαση συμπροεδρεύουν ε, οι πρόεδροι των δύο επιτροπών, Λίμπε και Αύκο, ο πρόεδρος Ταγιάννη και εγώ, και είμαστε υποχρεωμένοι να Είμαστε αυστηροί στην τήρηση του χρόνου. Υπάρχει χρονοδιάγραμμα για την αίθουσα, για τη διερμηνία ε, και για να υπάρχει και σεβασμός. Παρακαλώ να είστε σύντομοι στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις σας για να τηρούμε τους χρόνους μας και να μην χρειάζεται να σας διακόπτω ούτε εγώ το πρόεδρος Σταγιάννη. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για τη συμμετοχή της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ Ελευθεριών. Είναι παλιά γνώριμη για μας η Επίτροπος Γιουροβά. Την τελευταία πενταετία τη συναντούσαμε. Έχει εμπειρία ως μέλος του Σώματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου κατήχει το χαρτοφυλάκιο για την δικαιοσύνη και την προστασία των καταναλωτών. Τώρα θα μας μιλήσει για τις αξίες και τη διαφάνεια. Και έχει και το συνορισμό και την καθοδήγηση. Και με άλλους επιτρόπους. Τον Τιτιέ Ρέντερ της δικαιοσύνης και της, η Έλενα ε, Γκάλη, Ντάλι μάλλον, για την ε, ισότητα. Το χαρτοφυλάκιο της κυρίας Γιώροβα καλύπτει τομείς πάρα πολύ σημαντικούς για την Επιτροπή μας θα πρέπει να συντονίζει τη διατήρηση του κράτους δικαίου, παρακαλώ, και δημοκρατία και μηχανισμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Επίσης, την πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσχώρηση στο ε, χάρτη θεμελιδών ε, δικαιωμάτων που τέθηκε σε ισχύ με τη Συνδίκη της Λισαβόνας πριν από 10 χρόνια. Επίσης την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ε, ψευδών ειδήσεων και τη διαφύλαξη της ελευθερίας, της έκφρασης, της ελευθεροτυπίας και της πολυφωνίας των μέσων ενημέρωσης. Όλα αυτά εγγράφονται στο θεματολόγιο αυτού του χαρτοφυλακίου και είναι ιδιαίτερα προσφυλή θέματα για μας και, και μας απασχολούν μεταξύ πολλών άλλων στις εργασίες μας στην Επιτροπή Ελευθεριών. Θα ακούσουμε πολύ μεγάλη προσοχή όσα θα μας πει η υποψήφια αντιπρόεδρος Ιούροβα σε αυτούς τους τόσο βασικού τομείς για την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα δώσω αμέσως το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων που συμπροεδρεύει, τον κύριο Ταγιάννη, για να κάνει τα εισαγωγικά του σχόλια. Κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ, να καλωσορίσω την υποψήφια την πρόεδρο Γιούροβα, να υπενθυμίσω ότι το βιογραφικό της και οι απαντήσεις στις γραπτές ερωτήσεις έχουν διανεμηθεί σε όλους τους βουλευτές και έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσω ότι η διάρκεια της ακρόασης είναι τρει ώρες και Χαίρομαι διότι το χαρτοφυλάκιο της Αντιπροέδρου περιλαμβάνει και τη διαμεσολάβηση μεταξύ ε, Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ε, ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σύστημα του Speech and Candidate, του επικεφαλής υποψηφίου και τις σχέσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Είναι ένα από τα πράγματα, πράγματα που θα αναλάβει εάν επιβεβαιωθεί η αντιπρόεδρια τη. Η αντιπρόεδρο θα εκπροσωπήσει επίση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη για τα θέματα αυτά ακριβώς. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη τροποποίηση του εκλογικού νόμου και να εξασφαλίσει και τη συμφωνία με το Συμβούλιο. Η υποψήφια αντιπρόεδρος θα πρέπει να υποστηρίξει τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το θέμα αυτό για να ενισχύσουμε τη διασυνοριακή διάσταση των ευρωεκλογών και έτσι να υπάρχει και δημοκρατική νομιμοποίηση τη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι στο χαρτοφυλάκιο της κυρίας Γιούροβα περιλαμβάνονται και η βελτίωση της λειτουργίας της πρωτοβουλία ε, των πολιτών και είμαι βέβαιος ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για την ε, ουσιαστική ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψη αποφάσεων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις γραπτέ, τη απαντήσει, είπε ότι θέλει να προχωρήσει πολύ σημαντικά θέματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για την Επιτροπή μας, όπως για παράδειγμα η επικύρωση του εκλογικού νόμου, το Μητρό Διαφάνειας επίσης. Ελπίζω να αποδειχθεί σημαντικό σύμμαχο ε, στην επόμενη πενταετία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως υπενθύμησε ο πρόεδρος ε, Λόπεθ Αγγιλάρ και επιτρέψτε μου να το επισημάνω και εγώ ως δημοσιογράφος, ένα από τα θέματα που θα πρέπει να συζητήσει είναι η ελευθεροτυπία, η ελευθεροτυπία των μέσων ενημέρωσης και Έχουμε ε, εντό ολίγου την επέτειο της τηλεφωνίας της ε, Καρουάνα Γκαλίτσια στη Μάλτα. Θα ήθελα λοιπόν να θυμηθούμε την ε, Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια και μαζί του θυμόμαστε και όλου του δημοσιογράφου που υπήρξαν θύματα στη μάχη που έδιναν για την αλήθεια. Και θα θέλαμε η μάχη για την αλήθεια για τη δολοφονία της Ντάφνη Καρουάλινα Γκαλότσο όπως και του Γιάνν Κούτζακ να λάμψει το συντομότερο δυνατόν. Πώς μπορούμε, κύριε Αντιπρόεδρε και αγαπητοί φίλοι, εμείς να ζητήσουμε από τη Ρωσία να εγγυηθεί την ε, ελεύθερη ενημέρωση και το σεβασμό των δημοσιογράφων. Πώς μπορούμε να ζητήσουμε από την Τουρκία να εγγυηθεί την ελευθερία ε, των δημοσιογράφων και την ελευθεροτυπία. Πράγματα τα οποία πρέπει να κάνουμε σε όλο τον κόσμο, εάν εμείς δεν είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των δημοσιογράφων. Να δώσω αμέσω το λόγο στην, αντιπρόεδρο, στην υποψήφια αντιπρόεδρο, την κυρία Γιούροβα. Έχετε 15 λεπτά στη διάθεσή σας. Αξιότιμα μέλη, κυρίες και κύριοι, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία να είμαι ξανά εδώ για την ακρόαση και να ζητώ και πάλι την εμπιστοσύνη σας. Επισκεπτόμουν συχνά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την τελευταία πενταετία και χαίρομαι που βλέπω τόσες πολλές οικίες φυσιογνωμίες. Προσβλέπω στη συνεργασία με όλους εσάς τα επόμενα χρόνια. Ο ρόλος μου στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν επιβεβαιωθώ από εσά, θα είναι να ασχοληθώ με κρίσιμα και λεπτά ζητήματα. Το χαρτοφυλόκιο αυτό είναι αυτό το οποίο θα μπορούσα να αποκαλέσω η ψυχή της Ευρώπης. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αφορά τους Ευρωπαίους. Όπως είπε και η μέλουσα πρόεδρος, το χαρτοφυλάκιο αυτό είναι απάντηση στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, είτε εσωτερικές είτε εξωτερικές. Ο στόχος μου λοιπόν θα είναι η Ευρώπη να γίνει πιο δημοκρατική και πιο διάφανη. Να είναι πιο ανθεκτική ενώπιον νέων απειλών και ψηφιακών και να είναι και πιο ικανή να αντιμετωπίσει τις αξίες που πρεσβεύουμε συμπεριλαμβανομένου και του κράτους δικαίου και της ελευθεροτυπίας. Όπως έγραψε και ο Τίμωθη Σνάιντερ, το Σύνταγμα αξίζει να το διασώσουμε. Το κράτος δικαίου αξίζει να το διασώσουμε. Ε, Τη δημοκρατία αξίζει να τη διασώσουμε. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα μπορούν και θα χαθούν εάν όλοι περιμένουμε να κάνει κάτι κάποιος άλλος. Το χαρτοφυλάκιο αυτό αποτελεί μαρτυρία ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα περιμένει και ξέρω ότι θα μπορέσω να βασιστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως έμπιστο σύμμαχό μου. Θα ήθελε επίση η Ευρώπη να γίνει πιο ισχυρή και πιο ενωμένη, δημιουργώντα ε, γέφυρες μεταξύ των διαφόρων πλευρών της ενωσή μας. Φέτο, στη Τσεχική Δημοκρατία, όπω και σε πολλέ χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, θα γιορτάσουμε την 30η επέτειο του τέλου ε, των ολοκληρωτικών καθεστώτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση του σήμερα έχει οικοδομηθεί στα ερήπια του τείχους του Βερολίνου, ε, στο πνεύμα του κινήματος της αλληλεγγύης του Σολιντάρκη στην Πολωνία, στην Βαλτική Οδό και στην Βελούδινη Επανάσταση στην πρώην Τσεχοσλοβακία. Εγώ έχω ζωηρές αναμνήσεις από εκείνες τις μέρες. Τις θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Επιθυμούσαμε αλλαγές, επιθυμήσαμε να ενταχθούμε στην ευρωπαϊκή κοινότητα όχι σε αναζήτηση υλικών αγαθών, αλλά σε αναζήτηση ελευθεριών. Οι ευρωπαϊκές αξίες είναι τα κοινά μας θεμέλια. Μας ενώνουν από το βορρά στο νότο, από την Ανατολή στη Δύση ξεπερνάμε τις διαφορές της γλώσσας, των πολιτισμών και των παραδόσεών μας. Γι' αυτό ακριβώς ε, το να τηρούμε τις αξίες μας, τα θεμελιώδη δικαιώματά μας, το κράτος δικαίου, πρέπει να είναι ο βασικός μας στόχος και θα πρέπει να αποτελεί και μοχλό της Ευρωπαϊκής Ενότητας και όχι ε, πηγή διχασμού. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα το οποίο θα ήθελα να τηρήσω στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ στις τρεις προτεραιότητές μου. Καταρχά, πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου με τον οποίο διορίζουμε και επιλέγουμε του Ευρωπαίου ηγέτε. Φέτο είχαμε αυξημένη συμμετοχή στι ευρωεκλογέ. Πρόκειται για μια ευκαιρία, καθώ επίση και ευθύνη. Δεν θα πρέπει λοιπόν να απογοητεύσουμε τι ελπίδε των πολιτών μα. Όπως δήλωσε η μέλουσα πρόεδρος, το πρώτο δίδαγμα είναι ότι πρέπει να βελτιώσουμε το σύστημα του κύριου υποψηφίου, αντιμετωπίζοντας και το θέμα των ε, ε, υπερεθνικών ε, καταλόγων, της υπερωθικής λίστας. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσω το ρόλο μου ως πρόεδρος ε, της ομάδας των επιτρόπων για μια νέα αίθουσα για την Ευρωπαϊκή δημοκρατία προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συμβάλλει ε, στις εργασίες της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης για τα θέματα αυτά. Για να είμαστε αξιόπιστοι και πλήρω υπόλογοι στα μάτια των πολιτών μα, πιστεύω ότι εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα θεσμικά όργανα πρέπει να αποτελούμε το υπόδειγμα. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι νομοθετικές διαδικασίες ε, θα είναι εύκολα αντιληπτές ε, και δεν θα υπάρχουν ε, κρυμμένα συμφέροντα. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να συνεργαστούμε για ένα μητρό διαφάνειας και ένα ανεξάρτητο σώμα δεοντολογίας, το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όπως προβλέπεται στις κατευθυντήρες γραμμές. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ ισχυρό σύμβολο τη αποφασιστικότητάς μας να βοηθήσουμε την Ευρωπαϊκή η πολιτική μας κουλτούρα και να σεβόμαστε τα υψηλότερα δεντολογικά πρότυπα. Δεύτερος πυλώνας της δουλειά μου θα ε, βασίζεται στο κράτος δικαίου και στην ελευθεροτυπία. Το κράτος δικαίου είναι η βάση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύη και της αμοιβέ εμπιστοσύνης. Είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για τη λειτουργία του ευρωπαϊκού δικαίου και της ενία αγοράς. Και ένα είναι βέβαιο. Δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι δεδομένο το κράτο δικαίου. Γι' αυτό ακριβώ θα πρέπει να υπάρχει μια νοοτροπία κράτου δικαίου που θα βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό. Θα πρέπει να προωθήσουμε το διάλογο και να αποφεύγουμε περιπτώσεις κρίσης. Αλλά θα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όταν προκύπτουν. Εγώ θα δρώ με αποφασιστικότητα αν χρειαστεί και θα χρησιμοποιώ όλα τα απαραίτητα εργαλεία. Όπως γνωρίζετε, ο Φραντ Τίμερμανς εργάστηκε κατάπαυστα στο θέμα αυτό και θεωρώ ότι εγώ θα συνεχίσω το έργο του στην επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν επιβεβαιωθώ, θα ε, συνεργαστώ με τον Επίτροπο Αρμόδιο για θέματα δικαιοσύνης για να ενισχύσουμε περαιτέρω την εργοθήκη για την αποτελεσματική ε, εφαρμογή του κράτους δικαίου και τον ετήσιο κανόνο της, ε, ε, του κύκλου της αναθεώρησης του δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει και ο Ευρωπαϊκός, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συζητήσει ένα μηχανισμό που εξετάζει την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και βασίζομαι σε εσά για να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τα επιτύχουμε αυτά με αποφασιστικότητα και δικαιοσύνη. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, η ψηφιοποίηση έχει επιφέρει πολλά ωφέλη και μπορεί να ενισχύσει τη δημοκρατία. Ωστόσο, έχει εκθέσει την ίδια τη δημοκρατία σε νέες απειλέ και έχει διευρύνει παλαιότερες απειλέ, συμπεριλαμβανόμενε τη εξωτερική παρέμβαση και της διάδοση παραπληροφόρησης και δεν είναι ίσονο σημασία σε αυτό το θέμα. Είναι πραγματική απειλή. Η πρόσφατη μελέτη της Οξφόρδης για την παγκόσμια τάξη παραπληροφόρησης βρήκε αποδείξεις για οργανωσμένες εκστρατείες χειραγώγησης μέσω των κοινωνικών μέσων σε 70 χώρες από τις 48 το 2018. Ε, δηλαδή ε, άνοδο ε, από τις 48 χώρες που είχαν διαπιστωθεί το 2018 σε ολόκληρο τον κόσμο υπάρχει μεγάλη προσπάθεια υποβάθμισης και υπόσκεψης της εμπιστοσύνης στη δημοκρατία. Όλα αυτά συμβάλλουν σε αυξημένη πόλωση στις κοινωνίες μας και αυτό μπορεί με τη σειρά του να οδηγήσει σε βία καθώς ε, σωματικές επιθέσεις ε, κατά των πολιτικών, των δημοσιογράφων ή μελών των μειονοτήτων συμβαίνουν και στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ε, το αγνοήσουμε. Οι εχθροί της δημοκρατίας έχουν χρησιμοποιήσει ήδη την σφαίρα, την ψηφιακή, σαν όπλο τους. Πρέπει να αυξήσουμε τις δυνατότητές μας να αντισταθούμε και να αντιδράσουμε. Ο Χάβελ ήδη είχε αντιληφθεί τις δημοκρατικές προκλήσεις όταν έγραψε στην προ-ιντερνετική εποχή και σας παραθέτω το φυσικό μειονέκτημα της δημοκρατίας είναι ότι εξαιρετικά κουραστική για αυτούς που την εννοούν, ενώ επιτρέπει σχεδόν οτιδήποτε, σχεδόν τα πάντα σε εκείνους που δεν την αντιλαμβάνονται σοβαρά. Και τέλος της παράθεσης. Και θέλω εγώ να προσθέσω κάτι. Σήμερα Θα ήθελα να προσθέσω το εξή και για αυτού που θέλουν να την καταχραστούν. Πράγματι, η περάσπιση τη δημοκρατία και των ελευθεριών δεν είναι εύκολο εγχείρημα και η εργασία μα δεν έχει ολοκληρωθεί. Είμαι αποφασισμένη να παγιώσω και να εδραιώσω αυτή μα την ανταπόκριση σε αυτή την απειλή, ενώ θα σέβομαι την ελευθερία λόγου. Και θέλω να τιμήσω όλου του συναδέλφου σε αυτήν την επιτροπή που εργάστηκαν επ' αυτού μαζί μου το 2018, ιδιαίτερα την είπατε εκπρόσωπο Μογκερίνη, τον αντιπρόεδρο Άνσιπ και την Επίτροπο Γκάμπριελ. Έχουμε κάνει κάποια σχετικά πρώτα αλλά είναι μόνο πρώτα Εάν με επιβεβαιώσετε, θα σχεδιάσω το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για τη Δημοκρατία, που η μέλουσα πρόεδρος έχει, μου έχει εμπιστευθεί και θεωρεί πως είναι ένα όχημα για να δοθεί μια νέα όθηση στην αντιμετώπιση αυτού του θέματος, ε, έτσι ώστε η δημοκρατία μας να είναι πιο ανθεκτική. Αυτό απαιτεί ένα ευφυές ρυθμιστικό πλαίσιο που να είναι συνεπέ ε, και να υπάρχουν διασυνδεδεμένες δομές. Θα εργαστώ επιλύσεων με μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική διαφήμιση και τη σαφήνεια ε, για τα οικονομικά των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων. Επίσης, ε, θα αξιολογήσουμε προσεκτικά κατά πόσο οι πλατφόρμες τηρούν τις υποχρεώσεις τους υπό τον κώδικα πρακτικής σχετικά με την παραπληροφόρηση. Αλλά χρειάζονται περισσότερα πράγματα. Χρειάζονται δυνατότητες και έρευνα για να μπορούμε να ανοιχνεύσουμε αντιμετωπίσουμε τις απειλές ε, νωρίτερα και καλύτερα σε επίπεδο κράτους μέλους. Επίσης, η κοινωνία να κατανοήσει το κλίμακα του κινδύνου και να βοηθήσουμε τον κόσμο να αυτοπροστατευτεί, αυξάνοντας τη γνώση, την ε, παιδεία, ιδιαίτερα την ψηφιακή ε, παιδεία. Έτσι λοιπόν για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την παραπληροφόρηση και για να οικοδομήσουμε την ανθεκτικότητα θα πρέπει να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση με ε, τις κυβερνήσεις, τα ενδιαφερόμενα μέρη, ε, τα πολιτικά κόμματα, τις πλατφόρμες, τους δημοσιογράφους, τους ερευνητές, ε, τους εκπαιδευτικούς και την κοινωνία των πολιτών. Και σε αυτό θέλω να είμαι σε στενό διάλογο μαζί σας και εκτιμώ ιδιαίτερα τη δική σας συμβουλή. Ένας άλλος τομέας εστιασμού θα είναι η ελευθεροτυπία και ο πλουραλισμός στα μέσα. Ε, και σίγουρα εδώ πιστεύω πως μπορούμε να κάνουμε περισσότερο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την χρηματοδότηση για ανεξάρτητα project που παρακολουθούν ε, ο πλουραλισμό στα μέσα, τι ε, παραβιάσεις στην ελευθερία του τύπου και την προστασία των δημοσιογράφων των οποίων η ασφάλεια κινδυνεύει. Εγώ θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσο που έχω στη δυνατότητά μου ώστε να προωθήσω τις εκθέσεις ε, της ε, ομάδας υψηλού επίπεδου. Τρίτος πυλώνας ε, το, τώρα των αρμοδιοτήτων μου είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι βασικά για να είναι η Ευρώπη ο χώρος που θέλουμε να, μένουμε. Ένταξη για όλους, ισότητα για όλους, ασφάλεια για όλους, ε, ε, ψηφιακή μεταρρύθμιση με επίκεντρο τον άνθρωπο. Γνωρίζω την ανάγκη να υπερασπίζομαι τους ανθρώπους και τα θεμελιώδη τους δικαιώματα καθημερινά, κάθε ώρα, κάθε λεπτό απειλούνται και δεν θέλουμε να αφήσουμε κανέναν ε, πίσω. Θα συνεχίσω την εργασία που ξεκίνησα υπό την σημερινή Κομισιόν για την προώθηση του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σύντομα θα γιορτάσουμε τη δέκατη επέτειο του χάρτη. Θα χρησιμοποιήσω εκείνη την επέτειο για να αναθεωρήσουμε τη στρατηγική μου. Η θέση μου ω Αντιπροέδρου, αν επιβεβαιωθώ, επιφέρει οριζόντια ευθύνη και θέλω να προωθήσω τα θεμελιώδη δικαιώματα σε όλα όσα κάνουμε. Θέλω τα θεμελιώδη δικαιώματα να το τοποθετηθούν στον, ε, στην αρχή στο σχεδιασμό της ε, χάραξης πολιτικής της Κομισιόν, είτε είναι για την τεχνητή νοημοσύνη, είτε πρόκειται για την ψηφιακή μετάβαση, είτε πρόκειται για τις πολιτικές ισότητας. Και θέλω να τονίσω το εξή. Τα θεμελιώδη δικαιώματα δεν αποτελούν εμπόδιο στην κοινοτομία. Αντιθέτως, μας βοηθούν να εξασφαλίσουμε πως οι λύσεις μας θα θέσουν τον άνθρωπο πρώτα και θα είναι πιο βιώσιμες ως αποτέλεσμα αυτού. Ας πούμε, θεωρώ, ε, ως παράδειγμα μάλλον, σημαντική πτυχή αυτού που θα κάνουμε στο μέλλον για τη στρατηγική μας, για την ε, ε, τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η προσέγγιση, είμαι πεπισμένη, θα μας τοποθετήσει σε ισχυρή θέση ως παγκόσμιους πρωτοπόρους που θεσπίζουν τις προδιαγραφές, όπως έχουμε κάνει εξάλλου και για την προστασία των δεδομένων. Τέλος, θέλω να εξασφαλίσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, έχει, θα, θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα είναι αυτό ένα πολύ ισχυρό μήνυμα στην προσήλωσή μα για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτέ, πιστεύω πω η Ευρώπη μπορεί να είναι ισχυρή και να προωθεί τι αξίε τη διεθνώ εάν είμαστε ενωμένοι. Χρειαζόμαστε καλύτερη και πιο και Ευρώπη και Ευρώπη με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση που να μπορεί να σταθεί για, ε, εξ ονόματος των πολιτών μας και να τους υπερασπίζει από τις παγκόσμιες απειλές. Και για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ενεργήσουμε καλύτερα από κοινού. Όλοι αυτοί οι τομεί βασίζονται ε, πολύ σε μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στην Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, θα επιτύχουμε αποτελέσματα με ισχυρή διαθεσμική συνεργασία. Θα είμαι πάντοτε έτοιμη να συνομιλήσω με το Κοινοβούλιο και τις Επιτροπές σας, ε, ιδιαίτερα σε όλα τα στάδια της χάραξης πολιτικής και της λήψης πολιτικών αποφάσεων μέσα από τον πολιτικό διάλογο στο πνεύμα πίστης, εμπιστοσύνης και πλήρους διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Για να ξεκινήσουμε καλά, σεβόμαστε και το χρονοδιάγραμμα. Πολύ καλό σημάδι. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Τώρα ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο τους επικεφαλής των πολιτικών ομάδων από την Επιτροπή ΑΦΚΟ και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Στη συνέχεια, μετά από τις πρώτες 7 ερωτήσεις και απαντήσεις, θα ξεκινήσουμε με το δεύτερο γύρο. Από τα μέλη της ε, ΑΦΚΟ, της Γιούρι, της ΛΥΜΠΕ. Πρώτος ομιλητής, η Ρομπέρτα Μέτσολα, συντονίστρια του ΕΛΚ στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία υποψήφια αντιπρόεδρε για την ε, εξαντλητική σας εισαγωγή και για την ε, προσήλωση που είχατε ως Επίτροπος την τελευταία αιτία. Σας έχει ανατεθεί ένα χαρτοφυλάκιο που είναι θεμελιώδης πυλώνας του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Αν επιτρέπουμε να απειλείται οπουδήποτε το κράτος δικαίου, κινδυνεύει να καταρρεύσει παντού. Έχουμε μακρά παράδοση στο Κοινοβούλιο με ένα μηχανισμό ε, ελέγχου σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα δεσμευτείτε να υπάρξει ένας τέτοιος μηχανισμός ε, και ακρογωνιός λήθος είναι η ελευθεροτυπία, όπως είπε και ο πρόεδρος Σταγιάννη στην εισαγωγή του. Τα τελευταία χρόνια είδαμε τις δολοφονίες των δύο δημοσιογράφων στη Μάλτα και τη Σλοβακία. Τι μπορείτε να κάνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε οι ε, δημοσιογράφοι να προστατεύονται όχι μόνο από τη δολοφονία στη ε, χειρότερη περίπτωση, αλλά από τη συνεχή παρενόχληση και τις διαδοχικές αγωγές και προσφυγές στη δικαιοσύνη και μηνύσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μετσόλα για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να ε, είμαι όσο γίνεται πιο συγκεκριμένη. Ε, λίγο προσωπικά, αν μου επιτρέπετε, σχόλια στην αρχή. Αναφερθήκατε στη δολοφονία της δάφνε Καρουάνα Γκαλίτσε και του Γιάν Κούτσιακ. Συναντήθηκα με την οικογένεια της Δάφνης στη Μάλτα. Είδα τη μητέρα της, τον πατέρα της και το γιο της και τους υποσχέθηκα, στη μητέρα της κυρίως, ότι θα παρακολουθώ πάρα πολύ στενά τις έρευνες που διεξάγονται σχετικά με τη δολοφονία αυτή. Γιατί η οικογένεια και η μητέρα της περιμένουν τη δικαιοσύνη. Και υποσχέθηκα και στο γιο της ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να προστατεύονται καλύτερα οι δημοσιογράφοι στην Ευρώπη, γιατί είναι και ο ίδιος δημοσιογράφος και πιστέψτε με, είμαι πολύ στρατευμένη σε αυτή την υπόθεση και σε αυτές τις υποσχέσεις. Και αν με επιβεβαιώσετε με πολύ μεγάλη χαρά θα κάνω περισσότερα για να τηρήσω αυτές τις υποσχέσεις μου και να εγγυηθώ καλύτερα ότι δεν θα υπάρξουν άλλες δολοφονίες δημοσιογράφων στην Ευρώπη. Το κράτος δικαίου και ελευθεροτυπία συνδέονται. η Ευρώπη δεν θα μπορούσε να λειτουργεί χωρί το κράτο δικαίου. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς να το διατυπώσω τώρα, είναι ένα συμβιβασμός που συνεχώς εξελίσσεται ε, πανευρωπαϊκά, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Υπήρου. Είμαστε καλοί στους συμβιβασμούς, αλλά θα πρέπει να είμαστε εξίσου καλοί ε, ε, στην αδιαλαξία όταν κάπου δεν θέλουμε να κάνουμε συμβιβασμούς γιατί δεν χωράνε συμβιβασμοί στο κράτος δικαίου, στην ε, ελευθερία για όλους και στην ισονομία για όλους. Και αυτή η αρχή του κράτους δικαίου χρειάζεται να προστατεύεται καλύτερα, να αντλήσουμε τα διδάγματά μας την τελευταία πενταετία είδαμε ότι θεωρούμε κάποια πράγματα δεδομένα που δεν ισχύουν. Χρειάζονται συνεχή διάλογο με τα κράτη-μέλη, συνεχή προσοχή και φροντίδα. Γιατί αν το κράτος δικαίου αποτύχει καταρρεύσει σε ένα-δύο κράτη-μέλη στην Ευρώπη, καταραίει και όλος ο χώρος ελευθερίας δικαιοσύνης για τη συκοφαντική δυσφήμιση ε, και τις ε, μηνύσεις που γίνονται κατά δημοσιογράφων για συκοφαντική δυσφήμιση. Υπάρχουν καταχρήσεις εκεί και θα πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται με το διεθνές ιδιωτικό δίκαιο. Μπορεί να χρειαστεί να ζητήσουμε κάποια νομική αρρωγή ε, ή και χρηματοδότηση ε, υπέρ των δημοσιογράφων που υφίστανται τέτοιες επιθέσεις. Συμπραγματική ερώτηση. Κάτι που ε, διερευνούσε η Δάφνη πριν δολοφονηθεί ήταν ε, η υπόθεση των διαβατηρίων που μπορούσε κανείς να αγοράσει ουσιαστικά, να δώσει κάποια χρήματα για να αποκτήσει ε, ευρωπαϊκή υπηκότητα. Υπάρχει εκεί διαφθορά, ε, θέματα διαπλοκής, πολιτικού χρήματος. Τα δικαιώματα λοιπόν των πολιτών έχουν να κάνουν με την ίδια την ταυτότητα της Ευρώπης. Δεν θα πρέπει ε, κάποιος πρωθυπουργός να μπορεί να ορίζει πόσο τιμάται αυτό το ευρωπαϊκό ε, διαβατήριο, αφήνοντα στην άκρη όλους του κατατρεγμένου και του απόκληρους που δεν έχουν τα χρήματα να τα πληρώσουν. Δεν έχει έρθει η ώρα να απαγορευτούν αυτά τα σχήματα. Συμφωνώ, αλλά δυστυχώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να το κάνει, δεν έχει την αρμοδιότητα να κάνει ένα τέτοιο νομικό βήμα. Ε, αυτό που έκανα εγώ ήταν μια πρόταση να είναι πιο διαφανές το σύστημα αυτό, αν θέλουν να το διατηρήσουν τα κράτη-μέλη και να έχουν περισσότερο έλεγχο για όλη τη διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχει σαφής απόδειξη ότι διαπλέκεται κάποιος. Δεν μπορεί κάποιο που έχει χρήματα να αγοράζει την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, την ηθαγένεια ενό κράτου μέλου, άρα και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται έλεγχος και δέουσα επιμέλεια ε, εκ των προτέρων να κατανοήσουμε ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να αγοράσουν το εισαγωγικών την ευρωπαϊκή ηθαγένεια, για ποιο λόγο και ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ότι το χρήμα αυτό δεν προέρχεται από παράνομες δραστηριότητες και δεν ξεπλένεται κτλ. θα συστήσουμε μια ομάδα εργασίας που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να έχουν πολύ καλύτερο έλεγχο ε, των καταστάσεων αυτών. Σας ευχαριστώ. Δεύτερος ομιλητής, η ομιλήτρια Γκαμπριέλε Μπίσοφ από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες Αντιπρόεδρος της ΑΦΚΟ. Κυρία Γιούροβα, στην επιστολή ε, για την εντολή σας αναφέρετε ότι θα έχετε αυξημένο ρόλο, ένα ρόλο διαμεσολάβησης Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τον κορυφαίο υποψήφιο, καντιντάτ και τα υπερεθνικά ψηφοδέλτια. Εδώ στο Κοινοβούλιο όλοι γνωρίζουν πόσο τιτάνιο είναι αυτό το έργο, Ηράκλειος Άθλος. Ε, στις γραπτές σας απαντήσεις... Ε, είδα λίγο να απαντάτε σε κάποια πράγματα, αλλά θέλω πιο συγκεκριμένα. Εσείς λέτε ότι θέλετε να αξιολογήσετε τις εμπειρίες. Ε, θέλω πιο συγκεκριμένα να μου απαντήσετε τώρα. Πώς το φαντάζεστε αυτό, ε, πώς θα δράσετε έτσι διαμεσολαβητικά. Έχετε κάποιες ιδέες πώς θα το προσεγγίσετε. Και επίση μας είπατε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλετε να συμμετέχετε ε, έτσι με ιδιαίτερο ρόλο και στην συγκεκριμένη διάσκεψη που θα γίνει για το μέλλον της Ευρώπης. Ε, μπορείτε λοιπόν να μας τα πείτε λίγο πιο αναλυτικά πώς ε, θα ενσαρκώσετε αυτό το ρόλο διαμεσολάβησης. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. φυσικά πραγματικά υπάρχει πολλή δουλειά εδώ και αυτό μου ανέθεσε η εκλεγμένη πρόεδρος έτσι ώστε κάθε φορά να κάνουμε μια δοκιμή, να αποτυχάνουμε και να ξανακάνουμε το ίδιο πείραμα μέχρι να πετύχει. Υπάρχει ε, το θέμα αυτό των υπερηθνικών ε, ψηφοδελτίων από το 1999 και του κορυφαίου υποψηφίου. Δεν έχω χρόνο για να σας κάνω την ιστορική αναδρομή γιατί με ρωτήσατε και για το μέλλον. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν σε αυτό το ρόλο. Συστήσαμε αυτή την ομάδα για τη διάσκεψη στο μέλλον της, για το μέλλον της Ευρώπης, να δούμε ε, ποιες είναι οι διάφορες πρωτοβουλίες και οι διάφορες επιλογές που έχουμε και για τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου και για τα υπερεθνικά ψηφοδελτία. Δεν θα πρέπει ε, να παραμελούμε και τη στάθμιση των ε, αριθμητικών στοιχείων δεν είναι καμία χώρα σε μια ονεκτική θέση και να μην κινδυνεύει η ισορροπία του εκλογικού συστήματος. Θα πρέπει να μελετήσω το εκλογικό σύστημα αυτό ε, ως προς το εφικτό, ε, τα θετικά και τα αρνητικά, τα συγκεκριμένα. Να σας αναφέρω ως θετικό θα μπορούσε ένα υπερεθνικό ψηφοδέλτιο να δώσει μια πιο ευρωπαϊκή διάσταση ή πιο ευρωπαϊκή προοπτική σε μια προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ, να μην αναλώνονται ε, ή να μην εστιάζουν στα εθνικά θέματα αυτές οι εκλογές, γιατί είναι ευρωπαϊκές εκλογές και για την Ευρώπη πρόκειται. Ένα από τα αρνητικά θα ήταν το εξή μετά τις εκλογές η εκλεγμένοι ε, βουλευτές θα πρέπει να παραμείνουν σε επαφή με την εκλογική τους περιφέρεια. Και όταν η εκλογική τους περιφέρεια είναι ολόκληρη Ευρώπη υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ε, και για το εκλογικό σύστημα θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί τώρα και να αναζητήσουμε εκείνη την λύση που προσφέρεται καλύτερα για να βελτιώσει την κατάσταση. Με ποια έννοια να αυξηθεί η δημοκρατική νομιμότητα και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ο κορυφαίος υποψήφιος, Spitzen candidate θα είναι ο υποψήφιος για τη θέση του Πρόεδρου τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κάνω ό,τι μπορώ. Στην αρχή έχουν το λόγο οι εμπειρογνώμονε και στη συνέχεια οι πολιτικοί. Νομίζω ότι είναι ρεαλιστικό το χρονοδιάγραμμα στα μέσα του 2020. Το καλοκαίρι θα έχουμε τις πρώτες προτάσεις. I am very sorry, but we need to... Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά θα πρέπει να σεβόμαστε το χρόνο μας, γιατί και μετά την ακρόασή μας ε, υπάρχουν και άλλες ακροάσεις. Ε, παρακαλώ, τηρείτε το χρόνο και εσείς παρακαλώ, κύριε Αντιπρόεδρε. Η κυρία Μπίσοφ, ε, Αντιπρόεδρος της ΑΦΚΟ. Δύο συμπροματικές πολύ μικρές ερωτήσεις. Έχετε ένα αγαπημένο μοντέλο για τη διαδικασία αυτή του κορυφαίου υποψηφίου Candidate γιατί είπατε ότι υπάρχουν διάφορα και θα θελήσετε να βελτιώσετε τη διοργανική συμφωνία σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Υπόσχομαι ότι θα τηρήσω τον χρόνο, θα φροντίσω να είναι όλο και πιο σύντομε οι απαντήσεις μου, γιατί ο χρόνος ε, περνάει. Ξεκινάω λοιπόν, γιατί ήταν πολύ σαφής η ερωτήση σας. Το αγαπημένο μου μοντέλο όχι, ακόμα δεν το έχω βρει. Πρέπει να μιλήσω με τις εμπειρογνώμονες, να δω τις επιλογές μου, να σταθμίσω τα υπέρ και τα κατά και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι ο προσανατολισμός μου είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα θέλω να είναι λαμπρό γιατί είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό για την Ευρώπη. Εάν ε, καταλήξουμε σε κάποια επιλογή θα πρέπει να είναι ε, στα μέτρα των πολιτών. Δεν θα είμαι συγκεκριμένη λοιπόν επ' αυτού. Όσον αφορά τη, τη Οργανική Συμφωνία, Πιστεύω ότι δεν εμπίπτει σε αυτό, αλλά θα πρέπει να δω ε, τι δυνατότητες υπάρχουν και να το συζητήσω και τον Μάρο Σεφτσοβιτς, ο οποίος είναι ε, αντιπρόεδρος, επιβεβαιώθηκε ήδη για τις διοργανικές σχέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τώρα η Άννα Τζούλια Ντόναθ από τη Λίμπε το Renew Europe. Έχετε το λόγο. Κύρια Επιτροπέ, αυτή τη στιγμή οι κυβερνήσεις της Ουγγαρίας και της Πολωνίας ε, βρίσκονται στη διαδικασία άρθρο 7 με ελάχιστα αποτελέσματα. Η διαφθορά συνεχίζεται σε πολύ μεγάλους ε, βαθμούς τι μπορείτε να κάνετε ώστε η Ουγγρική και η Πολωνική κυβέρνηση να σεβαστούν τους ίδιους κανόνες με όλους και τα δικαιώματα των Ούγγρων και Πολωνών πολιτών να προστατεύονται. Θα συνεχίσετε με την απόφαση του άρθρου 7 που ε, έλαβε το Κοινοβούλιο πέρσι. Ε, πιστεύετε ότι η παρούσα προσέγγιση Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αποτελεσματική. Συμφωνείτε ότι αυτό δίνει το πράσινο φω φως και σε άλλους ε, ενδυνάμει ε, ε, οπαδούς του ολοκληρωτισμού στην Ευρώπη και ότι αυτό δεν βοηθά σε καμία περίπτωση την Ευρώπη και τις υπόλοιπες κυβερνήσεις. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντόνατ. Ε, σαφέστατη η ερώτησή σας. Καταρχάς, όσον αφορά το κράτος δικαίου, εν γέννη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακα τη συνθήκη και πρέπει να παρακολουθούμε την κατάσταση σε όλα τα κράτη-μέλη και όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει συστηματική παραβίαση και αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό κάναμε με την περίπτωση τη Πολωνία. Επίση, συμμετείχαμε στη συζήτηση για το άρθρο 7 στο Συμβούλιο για τη χώρα σα, για την Ουγγαρία. Και δεν συμφωνώ ότι όλα αυτά έγιναν ε, για το τίποτα. Η διαδικασία του άρθρου 7 είναι κάτι το οποίο δεν πίστευα ποτέ ότι θα ενεργοποιήσαμε, αλλά υπάρχει αυτή τη στιγμή ενεργοποιημένη και υπάρχει μια συζήτηση ε, σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Οι χώρες θα πρέπει να πούν και αυτέ πώς βλέπουν την αρχή του κράτους δικαίου και πώς θα πρέπει να την ε, τηρούν ε, συγκεκριμένα στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Αυτή όμω δεν είναι η μόνη διαδικασία. Εμεί, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιούμε έχουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας και διαδικασίες επί παραβάση. Υπάρχουν αρκετές παραβιάσεις αυτή τη στιγμή, ε, διαδικασίες σε εξέλιξη για την Ουγγαρία και κάποιες εξ αυτών Εάν δεν καταλήξουμε σε κάποιο σωστό συμπέρασμα με την Ουγγαρία, μπορεί να καταλήξουμε στα δικαστήρια. Και εκεί θα είναι η πιο κρίσιμη στιγμή. Και μάλιστα και για την Πολωνία, και αυτό φυσικά ισχύει για όλες τις χώρες. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι η αρμόδια αρχή για την ερμηνεία του νόμου. Και όταν λαμβάνονται οι αποφάσεις, ε, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, ε, ουσιαστικά μας επιτρέπουν να προσπαθούμε να πείσουμε με περισσότερη ασφάλεια τα κράτη-μέλη ε, για τον νόμο και θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Μέχρι τώρα. Ελπίζω να ε, λειτουργήσει το σύστημα έτσι. Αυτό είναι ο σταθερός μας πυλώνας και θα πρέπει να συνεχιστεί η συζήτηση ε, για τη διαδικασία του άρθρου 7, αλλά θα συνεχίσουν και διαδικασίες επί παραβάση. Εμείς προτείνουμε το κράτος δικαίου να είναι και ένας από τους όρους για το νέο προϋπολογισμό. Θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε με δίκαιο και διάφορο τρόπο αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει και κάτι με βάση τον προπολογισμό, γιατί οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι περιμένουμε να ε, προστατεύσουμε καλύτερα τα χρήματά τους. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά από πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, κάποια ήδη τα κάνουμε και πιστεύω ότι μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε κάτι σωστό και επαναλαμβάνω υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και εκεί τα πράγματα φτάνουν στην κορύφωσή τους. είμαι βέβαιη ότι αν χρησιμοποιήσουμε με δίκιο τρόπο όλα τα εργαλεία στη διάθεσή μας, θα μπορέσουμε να ε, έχουμε κάποια πρόοδο. Είστε υποψήφια την πρόεδρος, αλλά σας παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο, λέει ο κύριος Σταγιάννη. Θέλετε να κάνετε περαιτέρω ερώτηση. Στι γραπτές σας απαντήσεις σα είπατε και συμφωνώ απολύτω, ότι το κράτο δικαίου είναι ε, άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Στην ακρόαση του, ο κ. Ρέιντερ επιβεβαίωσε ότι ο κύκλος ετήσιας ε, αναθεώρησης θα εξετάει κυρίως ε, την δικαστική ανεξαρτησία, την καταπολέμηση της ε, διαφθοράς, ε, τη δημοκρατία και τα μέσα ενημέρωσης. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι η ετήσια έκθεση θα καλύπτει και το πλήρη στόχο του άρθρου 7, δηλαδή και τα δικαιώματα ανεξάρτητων μη κυβερνητικών οργανώσεων και πολυφωνία των μέσων. Και επίση, μπορείτε να μα εγγυηθείτε ότι η ετήσια έκθεση θα περιλαμβάνει και συστάσει αναχώρα, όπω πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. μπορεί και εδώ να πρέπει να μακρηγορήσω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι πιο λακωνική. Όσον αφορά το νέο μηχανισμό που προτείνουμε, βάσει και των όσων πρότεινε το Κοινοβούλιο το 2016, βασιστήκαμε σε αυτό, πήραμε πολύ σημαντικά στοιχεία και σκέλη της πρότασης. Ε, ε, ζητάμε να υπάρχει ισορροπία εξουσιών που είναι κάτι το οποίο βρίσκεται υπό τη σκέπη του κράτους δικαίου και μάλιστα πολύ σαφώς. Και επίσης, ανεξαρτησία του δικαστικού, το δεύτερο θα είναι η διαφθορά και μετά ελευθεροτυπία και πολυφωνία των μέσων. Θα υπάρχει και μία άλλη σειρά θεμάτων όπου περιμένουμε να συνεργαστεί και στενά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί μας. Ε, η επικαιροποίηση της στρατηγικής για τα θεμελιώδη δικαιώματα θα είναι δύο παράλληλες διαδικασίες αυτές και θα υπάρχει και ένα σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία, ε, στο οποίο θα επισέλθουμε σε περισσότερο επίπεδο λεπτομέρειο όσον αφορά την πολυφωνία των μέσων, ε, την παραπληροφόρηση και την προστασία των εκλογών. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε τρία σκέλη στη δουλειά μας, ε, όπου θα υπάρχει ιδιαίτερα έντονη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Για τους πρασίνους τώρα, Τέρι Ρέντκε. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κυρία ε, Επίτροπε που ήρθατε. Και όντως ο, ο αγώνας για το κράτος δικαίου ε, συνεχίζεται και εκατομμύρια ε, Ευρωπαίοι περιμένουν να υπερασπίζεστε πάντα τα το άρθρο 2. Ε, τώρα, θέλω να μιλήσω για την κοινωνία των πολιτών και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω πως εδώ μπορεί να πέσουμε σε μια παγίδα. Από τη μια πλευρά δηλαδή να έχουμε μια διαδικασία για το κράτος δικαίου, και την αναθεώρηση, όπου συγκεντρώνουμε ενδιαφέρουσε πληροφορίε, αλλά δεν έχουμε απτά αποτελέσματα για τα κράτη-μέλη. Και από την άλλη να έχουμε το άρθρο 7, το, που όμω αυτή η διαδικασία εύκολα μπορεί να μπλοκαριστεί στο Συμβούλιο αν ένα κράτο μέλο διαφωνεί. Θέλω λοιπόν να σα ρωτήσω πώ θα εξασφαλίσετε πω αυτέ οι διαδικασίε θα συνδέονται σε ένα μέσο οικονομική κύρωση ε, σε περίπτωση που υπάρξουν παραβιάσει του κράτου δικαίου και πώ θα εξασφαλίσετε πω κάτι τέτοιο θα έχει απτέ επιπτώσεις για το εν λόγω κράτος μέλος. Δεν θέλω να μιλήσω για κυρώσεις, ε, θέλω να μιλήσω για σύνδεση ή για όρους ερεσιμότητα σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό και το κράτος δικαίου. Περισσότερο εννοούσα ένα σύστημα παρακολούθησης εκεί όπου θέλουμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ανα πάσα στιγμή ότι τα ότι θα προχωρήσουμε σε, στα κατάλληλα βήματα ε, σε σχέση με την παραβίαση αυτών των κανόνων που ισχύουν και θα εξετάσουμε όλα τα στοιχεία του συστήματος ε, και θα χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό που προβλέπεται στην πρόταση, δηλαδή στο πακέτο του δημοσιονομικού κανονισμού που θα ενεργοποιήθηκε σε περιπτώσεις περίπλοκες όπου θα βλέπουμε πραγματικά πως δεν υπάρχει έλεγχος ε, για τα χρήματα για το... ή ε, εκεί όπου διαπιστώνεται κατάχρηση. Δηλαδή δεν θα, το, δεν θα, δεν θα τιμωρηθεί ο δήμαρχος, η ΜΚΟ ή η, δικαιούχοι του συστήματος. Δεν είναι αυτός ο στόχος. Θέλουμε όμως οι κυβερνήσεις να είναι πιο, εύκολη, πιο δύσκολη ζωή τους όσον αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο. Και είμαι ευτυχής που η Φιλανδική Προεδρία ανακοινώνει πως υπάρχει όλο ένα και μεγαλύτερη στήριξη για αυτού του είδους την αιρεσιμότητα στις διαπραγματεύσεις για τον νέο προϋπολογισμό, διότι πιστεύω πως όντως μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο. Θέλετε να κάνετε περώτηση, μάλιστα. Μάλιστα, πρέπει να αντιδράσω. Ο συνάδελφο ε, ανέφερε τι ε, συνεχιζόμενε διαδικασίε κατά τη Ουγγαρία και τη Πολωνία υπό το άρθρο 7. Γνωρίζετε πω αυτή τη στιγμή ε, γίνεται μια πολιτική απόπειρα ώστε το Κοινοβούλιο να τεθεί εκτό αυτή τη διαδικασία. Εσεί θα είστε σύμμαχό μα ώστε να έχουμε ισχυρό ρόλο σε αυτέ τι διαδικασίε εφόσον είμαστε οι άμεσα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πολιτών. Και η δεύτερη μου ερώτηση είναι η εξή. Είπατε όταν ρωτηθήκατε για το πώ βλέπετε το ρόλο σας τα επόμενα πέντε χρόνια ότι δεν θα είστε μια δεύτερη Φραντ Τίμερμανς και ότι θα βρείτε το δικό σας στυλ. Πιστεύω πως εδώ όλοι μας ενδιαφερόμαστε για το ποιο θα είναι αυτό το στυλ και πώ θα διαφέρει από αυτό του Φραντ Τίμερμανς γιατί Πρέπει να ομολογήσω που, ότι ήμουν πολύ ικανοποιημένη που ο Φραν Τίμερμαν υπερασπίστηκε ενεργά και δραστήρια το κράτο δικαίου. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω και να δω πώ θα διαφοροποιηθείτε στο στυλ σα από εκείνον. Μάλιστα, ευχαριστώ για την επερώτησή σας, ε, κυρία Ρέτκε. Δεν μπορώ να φανταστώ πώ μπορεί να αποκλειστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τη διαδικασία του άρθρου 7, ενώ εκείνο είναι που την ενεργοποίησε αρχικά ε, Εάν θα είμαι δεύτερο, ένας δεύτερος streamer ε, έχω ε, κάνει πρόβες ε, πολλές φορές, γιατί οι δημοσιογράφοι με ρωτούν αν θα είμαι περισσότερο Timmermans ή λιγότερο Timmermans. Σίγουρα δεν είμαι Timmermans, αλλά όταν δύο άνθρωποι κάνουν το ίδιο πράγμα, ποτέ δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Πρέπει να πω ότι εγώ θαυμάζω τι έκανε ο Φραντς Τίμερμανς και το τι έχει επιτύχει. Δεν ήταν εύκολη δουλειά. Το να υπερασπίζεται κανείς το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι εύκολο καθόλου. Αλλά αυτό το κάνω όσο μπορώ καλύτερα κινητοποιώντας τη γνώση μου, την εμπειρία μου και από τις τοπικές, ε, την τοπική αυτοπεδιοίκηση που είχαμε προβλήματα, τις ικανότητες μου για διάλογο, αλλά θα είμαι αυστηρή όσον αφορά τις αρχές. Αυτό είναι σίγουρο. θεωρώ πως είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να διορθωθεί στην Ευρώπη και είμαι ευτυχής που με ανατέθη να εργαστώ για αυτό το ζήτημα μαζί με τον συνάδελφο Didier Renders. Και τώρα από την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία στη Λίμπε, ο κύριος Νίκολαους Φέστ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Έχει γίνει μια αλλαγή Ρινάλντι για λόγους ταξιδίου. Σας ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη και ε, κυρία υποψήφια επίτροπε κυρία Γιούραβα. Μεταξύ των υπολείπων καθηκόντων σας θα πρέπει να υπερασπιστείτε τον πλουραλισμό στα μέσα που είναι πυλώνας για τη δημοκρατία. Ας πούμε, στην Ιταλία έχουμε ένα κοινό πέντε φορές μεγαλύτερο, δηλαδή 24 εκατομμύρια κόσμο που, μετα... που ενημερώνεται μέσω των κοινωνικών μέσων, ενώ έχουμε και πολλά ε, έντυπα μέσα ακόμα. Τι εγγύηση θα δώσετε όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, αποφεύγοντας τα ιδιωτικά μέσα να εκφράζουν απόψεις οι οποίες μπορεί να επιβαρύνουν τη δημοσιογραφία. Ας πούμε, κόμματα τα οποία έχουν την άδεια να συμμετέχουν στις εκλογές, στην ουσία λογοκρίνονται. Το Κοινοβούλιο έχει κλείσει σελίδες ε, κινημάτων, πολιτικών κινημάτων, χωρίς να έχει ε, βγάλει τέτοια απόφαση η δικαιοσύνη. Τέτοια πράγματα περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης. Εσείς τι μέτρα προτίθεστε να λάβετε για να τα ε, αναγετήσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Ε, σας έχω καλά νέα. Δεν θα υπονομευθεί η ελευθερία του λόγου. Σίγουρα όχι από τα δικά μας σχέδια. Ε, δούμε τι γίνεται με τη δημοσιογραφία και το πώς μοιράζονται οι πληροφορίες. Έχουμε δημόσια μέσα ενημέρωσης, ανεξάρτητα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης στην ελεύθερη αγορά και μετά έχουμε και τα κοινωνικά μέσα και τις κοινωνικές δικτύωσης που αυξάνουν σε σημασία και σε όγκο στα κράτη-μέλη. Δείχνουν οι στατιστικές ότι τραβούν την προσοχή όλο και περισσότερο. Υπάρχουν κάποιες χώρες όπου ήδη ακούμε ότι ε, πάνω από τους μισούς πολίτες ενημερώνονται μόνο από το ίντερνετ και τα social media. Και αυτό έχει τεράστια επίπτωση ε, στη διαμόρφωση της κοινή γνώμης. Αυτό που θα κάνουμε όμως τώρα στο συγκεκριμένο τομέα, η ελευθερία της έκφρασης θα παραμείνει βασική ε, αρχή και αξία εξορισμού και είναι αδιαπραγμάτευτη, εκτός εάν το περιεχόμενο είναι παράνομο. Αυτό το κάνουμε για τη ρητορική μίσους, ας πούμε, στο διαδίκτυο. Δεν πρόκειται να προωθήσω καμία λύση ή καμία πρόταση που να προτείνει ότι ε, κάποιος θα πρέπει να είναι κριτής των όσων γράφονται στα μίδια. Δεν θα υπάρχει Υπουργείο Αλήθειας ούτε Επίτροπος Αλήθειας και τίποτα τέτοιο. Αυτό που θέλουμε όμως σε σχέση με τις κοινωνικές πλατφόρμες και τα social media είναι περισσότερη διαφάνεια. Εμείς δεν θα υπαγορεύσουμε τι θα πρέπει να διαβάζει ο κόσμος ή τι θα γράφει, αλλά θέλουμε οι πολίτες να γνωρίζουν την πηγή της πληροφορίας. Και όταν είναι πολιτική εκστρατεία, ποιος κρύβεται από πίσω και ποιος πληρώνει. Αυτό θέλουμε, περισσότερη διαφάνεια να επιτύχουμε για το συγκεκριμένο. Και ταυτόχρονα θέλουμε να έχουν περισσότερες ευθύνες οι κοινωνικές πλατφόρμες και να ε, αντιταχθούν ε, στα bots, ε, στην τεχνική, την νοημοσύνη και στους ψευδείς λογαριασμούς που διασπείρουν ψευδείς ειδήσει. Επίσης υπάρχει και το θέμα της ασφάλειας, αλλά μπορεί να επανέλθω στη συνέχεια. Θέλετε να απαντήσετε. Επομένως, εσείς συμφωνείτε ότι δεν θα αφήνετε πλέον σε ιδιώτες διαχειριστές ε, μέσω κοινωνικής δικτύωσης να καθορίζουν αυτά τα πράγματα. Λέτε ότι θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα είναι καθορισμένος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο οποίος θα είναι αρμόδιος για θέματα λογοκρισίας. Γιατί ουσιαστικά αυτά γίνονται καθαρά από ιδιωτικού ε, φορείς και δεν ξέρουμε τι απότερου στόχου έχουμε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που θέλουμε να κάνουν οι πλατφόρμες είναι το εξής να κοιτάνε τη ρητορική μίσους και τη ρητορική βίας ε, στο ίντερνετ και όταν ε, είναι ξεκάθαρο ότι κάποιος ε, υποδαβλίζει το, το, το μίσος και ε, καλεί κάποιον να προχωρήσει σε δολοφονία, ας πούμε, γιατί έχω δει στο Δουβλίνο, στα κεντρικά της Facebook, ε, τρομακτικά πράγματα να γράφονται, τότε η πλατφόρμα ε, πρέπει να επιλαμβάνεται, αλλιώς θα διαμαρτυρηθούμε. Αυτό θέλουμε να κάνουν, να σέβονται τον νόμο. Όταν ε, κάτι απαγορεύεται στη ζωή θα πρέπει να απαγορεύεται και στο ίντερνετ. Και δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση, εκτός αν θέλετε να έχετε εκατοντάδες χιλιάδες χωροφύλακες του διαδικτύου. Ε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλο η παραπληροφόρηση όμως. στο ποινικό δίκαιο δεν είναι παράνομο περιεχόμενο με την ποινική έννοια. Ε, εκεί θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο τι θέλουμε να κάνουμε και τι θέλουν να κάνουν οι πλατφόρμες. Αυτό θα κάνω. Ε, την ομάδα ECR, ο συντονιστής της ΑΦΚΟ, ο κύριος Χέρτ Κουρζουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, υποψήφια Αντιπρόεδρε. Σωστά είπατε ότι σας έχει αναθέσει η κυρία Φόντερ Λέιεν την υπεράσπιση και την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και του κράτους δικαίου. Είμαστε όλοι ενωμένοι στην πολυμορφία και έχουμε μία κοινή γλώσσα και είναι η γλώσσα του διαφωτισμού. Πλην όμως βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σηκώνει κεφάλι ε, η ανελευθερία, όχι μόνο εκτός της Ένωσης και εντός. Προηγουμένως είπατε ότι οι Τσέχοι συμπατριώτες σας ε, αναζητούσαν ελευθερία στην ένταξή σας στην ευρωπαϊκή κοινότητα τότε. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε όλα τα μέσα, είπατε, για να υπερασπιστείτε το κράτος δικαίου. Πολύ συγκεκριμένα, πώς το φαντάζεστε αυτό και μήπως χρειάζονται και επιπλέον συμπληρωματικά μέσα και εργαλεία να το κάνετε αυτό και ποια θα είναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπουρζουά για την ερώτησή σας. Πώς θα προασπίσω το κράτος δικαίου και μιλήσατε και για την ανελευθερία, η οποία πραγματικά αυξάνεται αυτό τον καιρό. Είμαι πεπισμένη ότι έχουμε ως σαφές κριτήριο της δημοκρατίας τις ελεύθερες εκλογές, έτσι, ή την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα βασικά. Ε, και γι' αυτό ε, μας θορυβεί ε, όταν βλέπουμε κάποιες εξελίξεις στα κράτη-μέλη ε, που ε, να απειλούν την ανεξαρτησία των ε, δικαστών προσπαθώ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν είναι δικηγόροι και νομικοί, που ευτυχώ δεν είναι όλος ο κόσμος δικηγόροι, ε, προσπαθώ να κάνω μία σύγκριση. Ότι όταν παίζει η ποδοσφαιρική σου ομάδα ε, και δεν υπάρχει ε, διαιτητής, πώς θα παίξει ποδόσφαιρο. Έτσι, διαιτητές στην κοινωνία είναι οι δικαστές. θα πρέπει ε, να δούμε ε, τις χώρες που υπάρχουν προβλήματα. Ήδη αναφέρθηκα στην προσφυγή επί παραβάση βάση του άρθρου 7 και τώρα είμαστε στη φάση της ε, συνολικής αξιολόγησης βάσει της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2016 για να έχουμε τη συνολική εικόνα, το πού βρισκόμαστε γιατί μας επικρίνουν ότι ε, χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, ε, ότι ε, καταφερόμαστε εναντίον συγκεκριμένων χωρών και μόνο ή τις κατατρέχουμε. Υπάρχουν και κάποια μέτρα προληπτικού χαρακτήρα και αυτή είναι η ετήσια επισκόπηση του κράτους δικαίου. Αυτό θέλουμε να λανσάρουμε και η πρώτη έκδοση θα έχει ολοκληρωθεί του χρόνου την Άνοιξη. Εκεί θα έχουμε την πλήρη εικόνα λοιπόν. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα πρόοδο. Και η συζήτηση για το κράτος δικαιού δεν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ στενή και να εστιάζει μόνο στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των θεσμών. Θέλουμε να δούμε και την ελευθεροτυπία και τη διαφθορά και ελπίζω αυτό να ε, φέρει καλά αποτελέσματα σε ένα σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Συμπληρωματική ερώτηση. Χωρίς μικρόφωνο, κύριε Μπουρζουά. Θα πρέπει να φροντίσουμε ε, να ζει το κράτος δικαίου ε, στα κράτη-μέλη, αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου στην ε, υπόθεση Αρανιώζη. Ότι όταν ζητείται η έκδοση ε, κάποιου ε, ε, να μην παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Στην αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης συμφωνείται να υπάρχει πάντα έλεγχος ως προς το εάν τηρούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γιατί ο χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων τώρα πλέον είναι πρωτογενές δίκαιο και κυριαρχεί ε, επί οποιοδήποτε άλλου δικαίου. Και μάλιστα αυτά τα λέει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στην ομολογία του. Συμφωνείτε και θα φροντίσετε αυτά να τηρούνται. Απάντης. Η υπόθεση Αρανιώση και κάποιες άλλες δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικός ο λόγος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και είναι πολύ ε, μεγάλη όθηση αυτή τα κράτη-μέλη όπου υπάρχει πρόβλημα. Πραγματικά το δείξατε κι εσείς ότι θα πρέπει να ισχύουν όλες οι αρχές και να προστατεύονται με τον ίδιο τρόπο και τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Αλλιώς η ευρωπαϊκή δικαστική συνεργασία δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσει και το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι τόσο επιτυχημένο εργαλείο στη δικαστική συνεργασία ε, που θα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα εάν παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα. Και αυτό είναι αντικείμενο του συναδέλφου Didier Reinders. Δεν θα αναθεωρήσουμε το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, θα μελετήσουμε ε, πώς λειτουργεί, θα το αξιολογήσουμε και ε, σε πρακτικό επίπεδο να δούμε ποιο ε, είναι το επίπεδο των φυλακών. Εγώ πρόσφερα στα κράτη-μέλη ενημέρωση και συμβουλές για τον, ε, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να αναβαθμιστούν ε, οι φυλακές. εξελίσσεται αυτή η προσπάθεια, συνεχίζεται, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως. Ευχαριστώ. Για να είμαστε σαφείς, ένα λεπτό για την ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση, ένα λεπτό για την συμπληρωματική ερώτηση και ένα λεπτό για την δεύτερη απάντηση. Να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ανσοφή Πελετιέ από την ΓΚΟΕ e και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε. Κυρία Επίτροπε, καλημέρα σας. Στην Ιπαλία, στην Ουγγαρία και στην Ιταλία εγκρίθηκαν ε, νομοθεσίες οι οποίες ε, παραβιάζουν το δικαίωμα των δημόσιων διαδηλώσεων. Και είχαμε και βία περιστατικά από πλευράς αστυνομία ε, στην Ισπανία και στη Ρουμανία. Και ως Γαλλίδα πολίτης αντιμετωπίζω και εγώ αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν λοιπόν θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία είναι ιερά στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής ε- Ένωσης και ο τα μέτρα για να πατάξουμε την αστυνομική βία δεν αρκούν. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω σκέφτομαι όλους εκείνους τους πολίτες που υπήρξαν θύματα αυτών των βιωτήτων όπως για παράδειγμα τα κίτρινα γυλαίκα στην ε, Γαλλία, τους δημοσιογράφους ε, και δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν τη δουλειά τους και διαδηλώσεις στους δρόμους που οι ε, αστυνομικές δυνάμεις ε, παραβίασαν ε, συνδικαλιστές, προσπιστές των περιβαλλοντικών δικαιωμάτων. Κυρία Επίτροπε, λοιπόν, ως αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια, πώς σκοπεύετε να εγγύθετε αυτά τα δικαιώματα στην δημόσια διαμαρτυρία, τα οποία είναι αδιαμφισβήτητα. Ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και η ελευθερία του συνέρχεσαι είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες την οποία πρέπει να προστατεύουμε και πάντα εξετάζουμε την κατάσταση στα κράτη-μέλη όταν υπάρχουν παρόμοια περιστατικά. Και όταν υπάρχει ανάγκη ε, γίνεται και συζήτηση με το κράτος μέλος. Σε αυτές τις συγκεκριμένες περιπτώσεις όμως εγώ δεν συμμετείχα σε αυτές τις συζητήσεις, ε, διότι ήταν ε, περισσότερο αρμοδιότητα του αρμόδιου επιτρόπου για θέματα ασφαλείας, ε, διότι αυτό είναι και θέμα ασφαλείας μεταξύ άλλων. Αυτό λοιπόν είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε μαζί με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια όταν θέλει κάποιο να ασκήσει το δικαίωμα τη ελευθερία του συνέρχεστε. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θέλετε να κάνετε συμπληρωματική ερώτηση. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα τώρα να σας ρωτήσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να διεξάγουν την αποστολή τους. Την προηγούμενη εβδομάδα, συνάδελφό σας, ο κύριος Ρέντερ, είπαν ότι η κατάρτιση είναι τρόπος ε, ώστε οι μη κυβερνητικέ οργανώσει να μπορέσουν να προχωρήσουν. Η, η πραγματικότητα όμω τελείω διαφορετική, κυρία ε, υποψήφια πρόεδρε. Το κράτο ε, δικαίου εδώ αυτή τη στιγμή ε, διακυβεύεται. Η κατάρτιση δεν αρχεί και δεν υπάρχει καμία αναφορά στο δημόσιο χώρο και στην ο διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Οι μη κυβερνητικέ οργανώσει δεν έχουν συνομιληθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχουν εκστρατείε δυσφήμιση και υπάρχουν και προβλήματα χρηματοδότηση. Κυρία Επίτροπε, την προηγούμενη εβδομάδα ακούσαμε την Καρόλα Ρακέτε, την οποία προσέβελαν στην Επιτροπή Λίντε κάποιοι συνάδελφοι και εδώ ε, πρόκειται και για ποινικοποίηση πάλι των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν σε ποιου ε, μπορούν να απευθυνθούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, τη σήμερα ημέρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν τους επιτίθεται. Θα κάνετε κάτι για να αλλάξετε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι εγώ ήμουν ο άνθρωπος ε, με τον οποίο πρέπει να έρθω σε επαφή στην παρούσα μου θέση αυτή τη στιγμή. Ήρθα σε επαφή με μη κυβερνητικέ οργανώσεις σε κάποια κράτη-μέλη και δεν ήταν καθόλου θετικά τα πράγματα, διότι η συζήτηση αφορούσε το γεγονό ότι δεν του έδιναν χώρο, δυσκολευόντουσαν συνέχεια οι συνθήκε εργασίες τους, προβλήματα λόγω αλλαγών στην νομοθεσία που του περιόριζαν επίση. Επομένω, θα ήθελα να συνεχίσω να είμαι ο άνθρωπο με τον οποίο θα έρχονται σε επαφή. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, κυρίω για μη κυβερνητικέ οργανώσει που δραστηριοποιούνται σε κοινωνικά εκεί εργασία, θα υπάρχουν κονδύλια στο Ευρωπαϊκό Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από, για πάρα πολλά χρήσιμα ε, προγράμματα και υπάρχει και το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας των Αξιών και των Δικαιωμάτων. Ο τρόπος με τον οποίο διαρθρώνεται για την επόμενη επταετία θα είναι ένα πολύ χρήσιμο μέσο χρηματοδότησης για να βοηθήσει όχι μόνο τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αλλά και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στα θέματα κοινωνικής εργασίας αλλά και στον τομέα θεμελιωδών δικαιωμάτων και ισότητας ενώπιον του νόμου, ε, ισότητα ενώπιον φορέων κλπ. Ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται ο πρώτος γύρος των ερωτήσεων και τώρα θα ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Ντανούτα Χούμπνερ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Αντιπρόεδρε, από το 2011 υπάρχει μια διοργανική συμφωνία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τα Μητρά διαφάνειας. Υπάρχει μητρό για τα λόμπι, υπάρχει και μια κοινή γραμματεία την οποία, η οποία εδράζει εδώ στο Κοινοβούλιο. Υπάρχει κώδικας διοντολογίας και ένα σωρό άλλοι κανόνες. Το, το Δεκέμβριο του 2016 η Κομισιόν αποφάσισε να υποβάλει μια νέα και διορθωμένη πρόταση για τη Οργανική Συμφωνία και συμφωνούσαμε συμφωνήσαμε με το Συμβούλιο πως οι τρεις θεσμοί θα ε, λειτουργούσαν με βάση αυτή τη συμφωνία. Πολλά είχαν επιτευχθεί και μετά η Κομισιόν έχασε το ενδιαφέρον της στη συνέχιση των διαπραγματεύσεων και αποχώρησε από τη Διαπραγματευτική Τράπεζα παρά την ισχυρή δεσμευσή του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση ε, αναστολής αυτών των διαπραγματεύσεων. Θέλω να δω, έχετε εσείς ε, βούληση να ξαναρχίσετε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Ε, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Χούμπνερ. Μπορώ να σας επιβεβαιώσω ναι, ότι με ενδιαφέρει πολύ το ζήτημα αυτό, όχι μόνο ως ε, επειδή υπάρχει στην εντολή μου, αλλά ε, νομίζω πως θα πρέπει να ξαναρχίσουμε το διάλογο ανάμεσα στους θεσμούς, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ άλλων για το Μητρό των Ομάδων Πίεσης και πώς χρησιμοποιούμε, αν είναι υποχρεωτικό ή εθελοντικό, και το δεύτερο ζήτημα είναι η πρόσβαση στα έγγραφα και το τρίτο είναι πώς θα μπορούμε να εγγυηθούμε ότι σε κάθε φάση της νομοθετικής διαδικασίας υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε αυτά που κάνουμε και στο διαδικασία που ακολουθούμε. Εγώ είμαι πεπισμένη πως ο κόσμος έχει το δικαίωμα να γνωρίζει τι κάνουμε και τι σχεδιάζουμε. Και στις περισσότερες περιπτώσεις τα αποτελέσματα των εργασιών μας οδηγούν σε περισσότερες υποχρεώσεις για κάποια τμήματα της κοινωνίας για τους πολίτες. Είναι σοβαρά πράγματα και πρέπει όσο γίνεται να ε, ε, γνωστοποιούμε και να κοινοποιούμε αυτά που κάνουμε. Τώρα, όσον αφορά το Μητρό Διαφάνειας, υπάρχουν τώρα 12.000 ε, καταγεγραμμένα άτομα και θεσμοί η Κομισιόν μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα παράδειγμα ότι δεν υπάρχει καμία συνεδρίαση χωρίς να καταγραφεί στο Μητρό και Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή το Κοινοβούλιο να το εξετάσει αυτό το θέμα με πλήρη σεβασμό στην ελευθερία εντολής. Δηλαδή εδώ δεν μιλάμε για επικοινωνία με τις περιφέρειες και τους ψηφοφόρους, αλλά μιλάμε για την επικοινωνία με τα λόμπι δεν έχω τίποτα εναντίον των λόμπι, αλλά ξέρουμε όλοι ότι εκπροσωπούν τα συμφέροντα άλλων. Άρα θα πρέπει να είμαστε διαφανείς για το πότε το συναντάμε και το τι κάνουμε. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε τη δυνατότητα βελτίωσης της πρόσβασης επί τη βάση της πρότασης του Ombudsman ε, εμένα μου αρέσει η πρόταση αυτή και πρέπει να επανέλθουμε και ξέρω πως υπάρχει σχετική συζήτηση στο Συμβούλιο όπου μιλούν για την εξισορρόπηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των διαπραγματεύσεων. Σωστό αυτό, γιατί πρέπει να το δούμε και από αυτή την άποψη. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα που θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να συζητηθούν σε έναν νέο διάλογο. Όσον αφορά την νομοθετική διαδικασία, το ίδιο ισχύει. Θα πρέπει να εξετάσουμε όλα τα στάδια και να δούμε και τη διαδικασία επιτροπολογίας. Ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε περώτηση. Μάλιστα, το Ευρωκοινοβούλιο είναι μάλλον το μόνο Ευρωκοινοβούλιο στο δημοκρατικό κόσμο που δεν έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας και η κυρία Βαντερ έδειξε ότι θέλει να προχωρήσει σε αυτό. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι πώς το βλέπετε εσείς αυτό το δικαίωμα πρωτοβουλίας για το Ευρωκοινοβούλιο γιατί πιστεύουμε πως επειδή εκλεγόμαστε άμεσα είναι σημαντικό στοιχείο για τη δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την ερώτηση, τη δεύτερη ερώτηση. Πιστεύω πως η υποψήφια πρόεδρος έχει στείλει ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς το Ευρωκοινοβούλιο γιατί είπε ότι θέλει να στηρίξει το δικαίωμα πρωτοβουλίας για το Ευρωκοινοβούλιο όταν ενεργεί με την πλειοψηφία των μελών της για τα ψηφίσματα μπορεί, να μπορεί δηλαδή να υιοθετήσει ψήφισμα που να ζητά υποβολή πρόταση από την Κομισιόν. Βέβαια σε αυτά σε πλήρη σεβασμό της ε, αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Αυτή είναι η επίσημη απάντηση που είναι απόλυτα σύμμορφη με την ανακοίνωση της υποψήφιας Προέδρου. Ναι, είμαι έτοιμη να το στηρίξω αυτή τη διαδικασία. Γιατί θα πρέπει να πω ότι στη διάρκεια της τρέχουσας εντολής μου Είχα ανέκαθεν σημαντική επικοινωνία με το Κοινοβούλιο, που ήταν όμως πάνω κάτω άτυπη. Ε, πήρα πολλές καλές ιδέες και προτάσεις από τα μέλη του Κοινοβουλίου. Μπορώ να πω ότι με βοηθήσατε, αλλά βλέπω πως το Κοινοβούλιο, καταλαβαίνω το, πως το Κοινοβούλιο θέλει όλα αυτά να οριστούν σε μια επίσημη και τυπική διαδικασία και ε, θα ε, εργαστώ με βάση τα όσα υποσχέθηκε η υποψήφια πρόεδρος. Και τώρα η κυρία Γκραπίνη των Σοσιαλιστών ΑΦΚΟ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, υποψήφια Αντιπρόεδρε, σας εύχομαι καλή τύχη πρώτα απ' όλα Μπορεί να απαντήσατε γραπτός και σήμερα προφορικά σε κάτι στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω. Αυτό είναι η εδραίωση της δημοκρατίας και η διαφάνεια που αναφέρεται και στην επιστολή ανάθεσης ε, της εντολής σας. Εσείς, ε, αν επιβεβαιωθείτε ε, ως αντιπρόεδρος, τι θα κάνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε να βελτιώσετε το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εφαρμογή μέτρων διαφάνειας για όλα τα θεσμικά όργανα, αλλά μέτρων φιλόδοξων εννοώ. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα έτσι ώστε να γίνονται σεβαστές οι κοινέ αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ανακτηθεί και να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκραπίνη. Πιστεύω ότι η ε, Επιτροπή δίνει το καλό παράδειγμα ε, έχουμε πάρα πολύ αυστηρούς κανόνες για τη διαφάνεια και δεν μιλώ μόνο ε, για το υποχρεωτικό μητρό διαφάνειας. Είναι και ο τρόπος με τον οποίο δημοσιεύουμε τα έγγραφα, με τον οποίο κάνουμε διαπραγματεύσεις. Είμαι πάρα πολύ περήφανη για τα όσα κάνει η Σεσίλια Μάνστρομ στις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο, καθώς επίσης και οι άλλοι συνάδελφοι στις διαπραγματεύσεις για το Brexit. Πραγματικά λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την υποχρέωση διαφάνειας που έχουμε και φαίνεται. Η ίδια μου η εμπειρία με το Μητρό Διαφάνειας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ξέρετε ότι χειρίστηκα πάρα πολύ δύσκολες περιπτώσεις Dieselgate, ε, προστασία προσωπικών δεδομένων που ήταν ε, ε, ολόκληρη ιστορία και ο ψηφιακό τομέα αντιδρούσε που είχαμε τόσους αυστηρούς κανόνες. Επίσης το ξέπλυμα χρήματος, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τρίτες χώρες. Άλλη μεγάλη ιστορία με τα λόμπι. Και αισθάνθηκα πολύ πιο ασφαλής και πιο ελεύθερη όταν ε, έπαιρνα αποφάσεις, ε, έχοντας πει ότι κοιτάξτε έχω συναντηθεί με τους μεν, με τους δε, όλα αυτά είναι στο Μητρό διαφάνεια τα έχω δηλώσει, ε, με ποιον συναντήθηκα, με ποιον μίλησα. Και πάντα το έκανα αυτό προς το, του συμφέροντος των Ευρωπαίων πολιτών. Έχουμε λοιπόν αυστηρούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα θέλαμε και τα άλλα θεσμικά όργανα να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό με πλήρη σεβασμό ότι σε κάστοτε ιδιαιτερότητας ε, και ανεξαρτησίας του θεσμικού οργάνου. Είναι πραγματικά σημαντικό να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτή την πορεία. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση? Ε, ε ακόμα και αν δεν μου είπατε τι θα κάνετε για να ε, επανέλθει ή να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Ένα τεστ ειλικρίνειας να κάνουμε. Συνεργαστήκαμε μαζί ε, στη θητεία σας αυτή την τρέχουσα που τελειώνει τώρα για την προστασία των καταναλωτών. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σας επιτυχία και ποια ήταν η μεγαλύτερη σας αποτυχία σε αυτόν τον τομέα. Ευχαριστώ. Well, thank you very much for this question. Uh, Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση αυτή. Θέλω να πω ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών αυξάνεται ακριβώς αυτό που κάνουμε τώρα, αυτό που συζητάμε, να λέμε τι κάνουμε, για ποιο λόγο το κάνουμε, ε, ότι συζητούμε με τους πολίτες κανονικά, δεν υπάρχουν κρυφές ατζέντε και κρυφά συμφέροντα, δεν κάνουμε ε, πολιτική έτσι και κλεισμένων των θυρών τύπου καμαρίλας και με ε, τρόπο ειλικρινή και ανοιχτό εργαζόμαστε και επικοινωνούμε για τους καταναλωτές. Υπάρχει μια νέα συμφωνία για τους καταναλωτές, οι συλλογικές αποζημιώσεις και οι αγωγές. Αυτό είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, που θα συνεισφέρει σημαντικά στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. Ό,τι κάνουμε στην καταπολέμηση του ξεπλήματος και της χρηματοδότησης της τριμοκρατίας επίσης είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα γιατί ε, τερματίσαμε κάποιες εγκληματικές πράξεις ε, βάλαμε ένα φρένο σε κάποιες πρακτικές. Έχουν γίνει πολλά. Παρ' όλα αυτά, ο Didier Renders έχει δουλίτσα μπροστά του ε, στη συγκεκριμένη ε, θητεία. Προστασία δεδομένων, ο κανονισμός τώρα είναι καθολικής αποδοχής και πρότυπο. Ευχαριστώ. Και τώρα ο συντηρητής της ομάδας New Europe από την Επιτροπή ΑΦΚΟ, ο κύριος Πασκάλ Ντουρά. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Γιούροπα και ευχαριστώ που ξεκινήσατε ε, με παράθεση του Βάλκλαφ ε, Χάβελ. Ε, χαίρομαι να ακούω να παρατίθενται τα λόγια αυτή τη μεγάλη προσωπικότητα. Τώρα, για να αντιδρώσω στα όσα είπε η κυρία Γκραπίνη, θα μπορούσε να μιλήσουμε και για τα όσα κάνατε για τα ε, σήματα εκτάκτου ανάγκη. Εγώ υπήρξα μάρτυρα. Δεν θα είχαμε μια τόσο αποτελεσματική οδηγία αν δεν είχατε μπλακεί εσεί με το θέμα αυτό. Μα είπατε όμω προηγουμένω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ο θεματοφύλακα των συνθήκων και πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ σημαντικό να το επενθυμίσουμε. Στην Επιτροπή ΑΦΚΟ υπάρχει μια δυσκολία που επαναλαμβάνεται για το θέμα της απαλλαγής του προπολογισμού του Συμβουλίου. Το γνωρίζετε. Εδώ και χρόνια προσπαθούμε να μας δώσει στοιχεία το Συμβούλιο για τη χρήση εκατομμυρίων ευρώ χονδρικά ε, τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες του. Η Επιτροπή του 2014 κάπου υπαναχώρησε και είπε ότι είναι θέμα μεταξύ Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εμείς ψηφίσαμε το 2016 κείμενο με το οποίο ζητούσαμε από το Συμβούλιο να μας δώσει στοιχεία και δεν το έκαναν. Κυρία Αντιπρόεδρε, λοιπόν, εσείς ε, βοηθήσατε θα βοηθήσετε το Κοινοβούλιο και τους πολίτες να μάθουν κάποια πράγματα και να υπάρξει κάποια διαφάνεια για τον προπολογισμό του Συμβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ντουράμ. Θα κάνω ό,τι μπορώ, διότι αυτό ήταν ε, στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας να κάνουμε πράγματα με μεγαλύτερη διαφάνεια που θα οδηγήσουν και αναπόφευκτα σε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη. Θα κάνω ό,τι μπορώ λοιπόν στον τομέα αυτό και φυσικά θα ζητήσω και τη συμβολή των εμπειρογνωμόνων μου, αλλά υπάρχει και η νομική ε, δυνατότητα που δίνεται στο Συμβούλιο να ε, δίνει τα στοιχεία του. Δεν γνωρίζω ακριβώς ε, τα στοιχεία, θα τα διαβάσω. Εάν δεν υπάρχει κάποιο νομικό πρόσκομα, δεν υπάρχει λόγος για τον οποίο το Συμβούλιο δεν θα πρέπει να δίνει τις πληροφορίες. Η απαλλαγή αφορά τεράστια κονδύλια και τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη. Επομένως, εγώ θα ήθελα να ζητήσω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια. Το μόνο που μπορώ να σας υποσχεθώ λοιπόν είναι ότι και επ' αυτού του θύματος ε, θα ε, είμαι αυτή η οποία θα βοηθήσει προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη διαφάνεια, παρά το γεγονός ότι ε, το Συμβούλιο είναι το αρμόδιο και πρέπει να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιορισμένες εξουσίες, ούτε καν εξουσία, μια κάποια ανεπίσημη πίεση θα μπορούσαμε να ασκήσουμε. Ευχαριστώ για τη βοήθεια και τα στοιχεία που μας είπατε για την οδηγία για τους ε, whistleblowers, ε, τους μάρτυρες ειδικού συμφέροντος, ε, σήμερα ψηφίζεται στο Συμβούλιο. Ήταν ένα από τα πολύ δύσκολα θέματα. Μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Και ίσως ελοχεύει ο κίνδυνο να δημιουργήσει και κάποιο χώρο για κατάχρηση. Υπήρχε πάντα το ερώτημα πώ θα διακρίνουμε τον καλό με τον κακό μάρτυρα δημοσίου συμφέροντο και πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε του σωστού διάβλους για να ενημερώσουμε για κάτι κακό. Ε, πρόκειται για ένα πάρα πολύ δύσκολο θέμα και ένα πολύ δύσκολο τριμερή διάλογο. Χάρη ε, στην πολύ ισχυρή δέσμευση του Κοινοβουλίου νομίζω ότι τα καταφέραμε και μπορέσαμε να έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ. Ο κύριος Ντουρά. Μια και το αναφέρετε, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο θέμα του τριμερούς διαλόγου. Μην σα πω ότι, θεωρήσετε ότι έχω θέματα εναντίον του Συμβουλίου, αλλά μια και το είπατε, ε, κάποιοι θεωρούν ότι ο τριμερής διάλογος είναι το μαύρο κουτί της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας ε, και ίσως να υφέρπει και μια κάποια αλήθεια εδώ. Πώς ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε τη διαφάνεια των τριμερών διαλόγων και των πληροφοριών από το Συμβούλιο που θέλουν από τη μια να έχουν τον τίτλο του συνομοθέτη και το δικαίωμα του συνομοθέτη επίσης, χωρίς όμως να ε, έχουν τις ίδιες συνθήκες και υποχρεώσεις διαφάνειας για τη δημοκρατία. Μπορείτε να μας πείτε δύο-τρία πράγματα λοιπόν για τα θέματα των τριμερών διαλόγων και αν ναι, ε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Καταρχάς, ε, και για τον τριμερή διάλογο, ιδιαίτερα για τον τριμερό διάλογο που είναι το τελευταίο στάδιο της έγκρισης της νομοθεσίας, θα πρέπει να υπάρχει όσο το δυνατό μεγαλύτερη διαφάνεια. Και πρέπει να σας πω ότι εγώ συμμετείχα σε πάρα πολλούς ε, τριμερείς διαλόγους και τον Ιούνιο αλλά και πριν. Και είναι εντυπωσιακό πόσο γρήγορα άλλαζε η πρόταση στα πλαίσια της διαδικασίας. Ορισμένες φορές είχαμε και δημιουργικές λύσεις επιτόπου και εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να δουλέψουμε. Γιατί πρέπει κάπως να βρεθεί συμβιβασμό. Πρέπει να επιτευχθεί ο συμβιβασμό και ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και εδώ είναι και η στιγμή όπου θα πρέπει να γνωστοποιούνται οι θέσεις των διαφόρων παικτών του παιχνιδιού θα εργαστούμε από αυτού, ε, θα δούμε και την πρόταση για τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, θα χρησιμοποιήσουμε την πρόταση της Φιλανδικής Προεδρίας που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και για τον τριμερή διάλογο και την πρόσβαση στα έγγραφα υπάρχει μια πολύ ζωντανή συζήτηση αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο και θα επανέλθουμε και στη συζήτηση για το πώς μπορεί να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια στους τριμερείς διαλόγους. Υπάρχουν παλιότερες προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πάλι να πω ότι πρέπει να αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια για να έχουμε ένα καλύτερο μοντέλο. Από την Επιτροπή Γιούρη, ο κύριος Γύρι Πόσπισιλ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αγαπητή κυρία Γιώροβα. Χαίρομαι πάρα πολύ που αναφέρετε το κράτος δικαίου επανειλημμένα στην εισαγωγή σας. Είναι αναπόσπαστο τμήμα του δικού σας χαρτοφυλακίου. Πιστεύω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι το ποινικό δίκαιο είναι στοιχείο του κράτους δικαίου. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να τιμωρείται μόνο ε, όταν ε, παραβιάζει τον νόμο και μόνο τότε όταν παραβαίνει ένα νόμο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το Γενάρη του 2018 ο Τσέχος Πρωθυπουργός, ο κύριος Μπάμπιτς, είπε ότι στην Τσεχική Δημοκρατία μπορεί να φυλακιστεί κάποιος ε, κατόπιν παραγγελίας και να προσαχθεί και στη δικαιοσύνη ε, ε, κατόπιν παραγγελίας. Συμφωνείτε με αυτά τα λόγια όταν θα αναλάβετε αρμόδια αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κράτος δικαίου πώς θα αντιδράτε όταν ακούτε τέτοια πράγματα από χίλιοι ηγετών για τη λειτουργία της δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. απάντηση. Θα απαντήσω ε, και εγώ ε, στα τσεχικά και σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ε, θα απαντήσω σε δύο σκέλη του ερωτήματος. Όπως γνωρίζετε, το 2006 υπήρξε πάλι ένα τέτοιο πολιτικό παιχνίδι. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλά, για το τι σημαίνει να σε διώκει μια πολιτική δικαιοσύνη που είναι στην υπηρεσία κάποιων πολιτικών και όχι του κράτους. Νομίζω όμως ότι από το 2006 η τσεχική δικαιοσύνη έχει διανύσει ένα πάρα πολύ μεγάλο δρόμο, έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Και είτε πρόκειται για πρωθυπουργό είτε για οποιονδήποτε άλλον. Όταν δηλώνουν ότι μπορούν κατά παραγγελία να διώκονται κάποιοι ποινικά, εγώ δεν το πιστεύω. Το αντίθετο, έχω πλήρη εμπιστοσύνη ε, στην ε, τσεχική εισαγγελία και στην τσεχική δικαιοσύνη. Είναι επαγγελματίες, αμερόληπτοι, ανεξάρτητοι και ε, διαδραματίζουν το ρόλο που τους αναλογεί σε ένα κράτος δικαίου. Ε, συμπληρωματική ερώτηση. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Αλλά θα μπορούσατε να απαντήσετε και στην άλλη ερώτηση που σας έκανα, που είναι πιο σημαντική. Δανείστηκα ως παράδειγμα μόνο την τσεχική δημοκρατία. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω, αν αναλάβετε αυτό το χαρτοφυλάκιο και επιβεβαιωθείτε ε, αρμόδια για το κράτος δικαίου στην Ευρώπη. Θα το θεωρήσετε ορθό όσο και απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή εσείς εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναλάβετε κάποια δράση, να αντιδράσετε σε τέτοια λόγια πολιτικών. Γιατί αυτά μπορεί να είναι εις βάρος του κράτους δικαίου. Εσείς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα πρέπει να αντιδρά ή απλώς να τα αγνοεί αυτά γιατί είναι τμήμα του πολιτικού παιχνιδιού. Απάντηση. Έχω ακούσει πάρα πολλές φρικτές ε, ιστορίες ε, και δηλώσεις από πολιτικούς στην Ευρώπη και πολύ συχνά ε, ήθελα να απαντήσω, αλλά δεν απαντούμε. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είμαστε θεματοφύλακες των συνθήκων και απαντούμε μόνο όταν υπάρχει κατά σύστημα ε, αλλαγή στους νόμους, στο κράτος δικαίου, κάτι που γίνεται ευνηδίως από τη μία μέρα στην άλλη και διακυβεύει ε, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Και είναι καλό θα έλεγα που δεν αναμειγνύεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε εσωτερικές υποθέσεις, ε, σχολιάζοντας δηλώσεις ε, έστω και ακραίες κάποιων εθνικών πολιτικών. Παρόλο που καμιά φορά θα ήθελα να μπορώ να αντιδράσω. Ο πρόεδρος της Επιτροπής LIBE, ο κύριος Λόπεθ ε, Αγγιλάρ. Κυρία υποψήφια Πρόεδρε Γιούροβα, είπατε την άποψή σα για το νέο όνομα και χαρτοφυλάκιο αξίε και διαφάνεια. Και πρέπει να σα πω δύο λόγια γιατί τα ονόματα έχουν σημασία, όπω είπε ο υποψήφιο αντιπρόεδρος κ. Χινάς όταν εξήγησε το όνομα του χαρτοφυλακίου του. Μα παρέπεψε στο William Shakespeare, στο όνομα του Ρόδου και μετά αναφέρθηκε και στον Ουμπέρτο Όκο, ο οποίο χρησιμοποίησε το όνομα του Ρόδου ω τίτλο σε ένα βιβλίο του. Ω ε, επίτροπος λοιπόν αρμόδια για τι αξίε και τη διαφάνεια θα πρέπει να πιέσετε για μια νέα ευρωπαϊκή δημοκρατία και θα συμμετέχετε και στη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη, πώ θα φροντίσετε η διάσκεψη αυτή να μην είναι μια διαδικασία ρουτίνα και να ε, προσεγγίσει τους Ευρωπαίους πολίτες, το κοινό και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών οι οποίες ε, συμμετέχουν στην όλη αυτή διαδικασία για το μέλλον της Ευρώπης και πώς θα δεσμευτείτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πάει πέραν της απλής υποστήριξης της ε, αξιολόγησης μεταξύ κρατών μελών και να υποστηρίξει την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρχουν ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, όπως γίνεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με την Επιτροπή της Βενετίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Φυσικά και έχουν ε, σημασία οι τίτλοι και τα ονόματα και για μένα είναι πολύ σημαντικό όμως και το χαρτοφυλάκιο όπως και το όνομα. Θα κάνω ό,τι μπορώ λοιπόν ώστε να του προσδώσω την κατάλληλη ουσία ώστε και οι πολίτες να καταλάβουν γιατί επικεντρωνόμαστε στις αξίες και στη διαφάνεια. Δεν είναι εύκολη αυτή η δουλειά, διότι οι αξίες είναι μια γενική αφηρημένη έννοια και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να είμαστε απόλυτα σαφείς ε, για τα σχέδιά μας και για αυτά που κάνουμε. Θα εργαστούμε σε τρεις πυλώνες όπως σας είπα. Ετήσια έκθεση για το κράτος δικαίου, όπου όπως είμαι βέβαιη ότι και ο Didier ε, θα προωθήσει τις ιδέες του για την αξιολόγηση μεταξύ κρατών μελών. Θα υπάρχει όμως μια αξιολόγηση που θα καλύπτει την ισορροπία την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του δικαστικού, τη διαφθορά και τα μέσα ενημέρωσης. Μετά θα έχουμε μια νέα όθηση για τη δημοκρατία που θα καλύπτει τις εκλογές, τον εκλογικό νόμο, την παραπληροφόρηση και πάλι θα έχουμε και την πολυφωνία των μέσων με ευρύτερο ε, πλαίσιο. Και το τρίτο το οποίο θα μας αποσχολήσει θα είναι η ε, στρατηγική για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Για μένα αυτά είναι η Αγία Τριάδα. Ε, η ελευθερία, τα θεμελιώδη δικαιώματα και η δημοκρατία και φυσικά εδώ θα θέλαμε και την ισχυρή δέσμευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, είμαι διατεθειμένη να κάνω την κατάλληλη παρακολούθηση και τη δουλειά εξορθολογισμού ώστε τα θεμελιώδη δικαιώματα να συμπεριληφθούν σε ό,τι κάνουμε, να λαμβάνουμε υπόψη τις αρχές αυτές. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εγώ δεν θέλω να βρεθώ πολύ ώρα στο γραφείο μου. Θέλω να είμαι έξω όσο περισσότερο γίνεται, σε συζητήσεις με τους πολίτες. Όχι μόνο με αυτούς οι οποίοι μας πιστεύουν. Ε, ξέρετε νομίζω όλη την κατάσταση, όταν οργανώνουμε μια διάσκεψη πάντα μιλούμε στους ίδιους και στους ίδιους και προσπαθούμε να πείσουμε αυτούς που ήδη ούτως ή άλλως μας πιστεύουν. Εγώ θέλω να πάω στα κράτη-μέλη, να μιλήσω στους φοιτητές και να κάνω πολύ περισσότερα προκειμένου να κατανοήσουν πολύ καλύτερα για ποιες αξίες δίνουμε αγώνα στην Ευρώπη. Επόμενη ερώτηση, κύριε Λόπεθ Αγγιλάρ. Ευχαριστώ και πάλι. Μία μικρή συμπληρωματική ερώτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στο χαρτοφυλακείο σας. Διεσμευόμαστε πλήρως ώστε να συμμορφώνονται όλοι προς το χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ακόμα και τα δικαιώματα των μειονοτήτων, που μπορεί να μην αρέσουν σε κάποιες κυβερνήσεις ή σε κάποια κράτη-μέλη κάποια στιγμή. Ε, κυρίως τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ, των Ρωμά, ε, μειονοτήτων, οποιασδήποτε μορφής, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι οι αξίες συνδέονται με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, που είναι και ο τίτλος του χαρτοφελοχείου του Αντιπρόεδρου Σχοινά για την εφαρμογή του άρθρου 2 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Εγώ δεσμεύομαι πλήρως να συνεχίσω αυτό που έκανα ούτως ή άλλως μέχρι τώρα να πω και πάλι ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, κυρίως την παρακολούθηση για τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εδώ αναφέρομαι στο χάρτη, αλλά και σε συγκεκριμένη νομοθεσία που αναφέρεται στην προστασία των μειονοτήτων και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων εν γέννη. Αυτό το οποίο έχω κατά νου είναι η απόφαση πλαίσιο για το ρατσισμό και την ξενοφοβία. Τα κράτη-μέλη υποτίθεται ότι θα έπρεπε να την εφαρμόσουν πριν από δύο χρόνια και αμέσω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να στέλνει επιστολέ, ε, διότι είδαμε ότι υπάρχουν κενά, έλλειψη συμμόρφωση, υπάρχουν κάποια κάποιες δυσκολίες, έλλειψη ενδιαφέροντος και σε κάποιες περιπτώσεις και ακόμα είμαστε στη διαδικασία και έχουμε και αρκετές διαδικασίες επί παραβάση οι οποίες έχουν ξεκινήσει. Το ίδιο και για την οδηγία για την ισότητα. Κάνουμε το, το ίδιο. Παρακολουθούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη και δεν παρακολουθούμε μόνο τη συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία που είναι και το βασικό μας έργο, αλλά προσπαθούμε να δούμε και πώς εφαρμόζονται στην πράξη οι νόμοι. Υποστηρίζουμε φορείς ισότητα στα κράτη-μέλη. Αυτή είναι βέβαια συμπληρωματική ερώτηση, οπότε δεν έχω χρόνο, ε. Ήθελα να πω και κάτι για τις φορείς της ισότητας, αλλά και αυτούς τους στηρίζουμε, να ξέρετε. Είμαι πολύ ευέλικτος, αλλά δεν ξέρω αν ο Λόπες Αγγιλάρ ε. είναι εξίσου κατά τη δική του τώρα προεδρία. Αναλαμβάνει λοιπόν τώρα την Προεδρία. Παίρνω το σφυράκι, παίρνω το σφυράκι. Daniel Freund τώρα, της ΑΦΚΟ. Ένα λεπτό. For answering our questions today. I'm over here. Um... Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι κάθε χρόνο χάνουμε από διαφθορά ε, το ισόποσο του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και βλέπουμε ότι η διαφθορά έχει φτάσει στα ύψη στα κλιμάκια και στη δική σας χώρα. Ε, δεν είδα όμως πουθενά τη λέξη διαφθορά διαβάζοντας τα χαρτοφυλάκια. Εσείς είπατε ότι θα επαγρυπνείτε για αυτό το θέμα και θα ήθελα παρακαλώ να το επιβεβαιώσετε. Σε αιτήσια βάση θα κοιτάτε τη κατάσταση της διαφθοράς και θα κάνετε συστάσεις στα κράτη-μέλη. Επίσης πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι αξιόπιστη ε, μπροστά σε αυτή τη μάχη κατά της διαφθοράς θα πρέπει να το αποδείξει. Όταν ε, ε, αποχώρησε, ε, αφιπηρέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μπαρόσο, η μισοί επιτροπή πήραν θέσεις σε λόμπι και υψηλόβαθμες και 24 φορές παραβιάστηκε το τελευταίο διάστημα ο κώδικας δεοντολογίας. Πώς θα εξασφαλίσετε λοιπόν και οι επίτροποι και οι ευρωβουλευτές δεν ε, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα κριτές και κρινόμενοι σε αυτά τα θέματα παραβίασης ε, ε, κωδικών δεοντολογίας. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φρόιντ. Καταρχάς γιατί τη διαφθορά. Όντως, αυτό που θέλουμε είναι να έχουμε μία ετήσια εκτίμηση της ε, διαφθοράς ε, στην ετήσια επισκόπηση του κράτους δικαίου. Γιατί εκεί ανήκει. Γιατί συχνά είναι ένα συνοδό φαινόμενο αυτό, ε, ένα επιφαινόμενο της φθήνουσας πορείας του κράτους δικαίου σε μια χώρα. Και όταν υπάρχει τέτοια φθηνούσα πορεία, η δικαιοσύνη και η εισαγγελία δεν αντιδρούν. Γιατί είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ψάρια για να διωχθούν. Βεβαίως ε, θα κοιτάξουμε με συστημικό τρόπο τη διαφθορά. Θα συνεχίσουμε. is Να κάνουμε τα εξής δύο. Και στο ευρωπαϊκό εξάμεινο Ε, επίσης, γιατί η διαφθορά ε, βλάπτει την οικονομία σε ε, ένα κράτος μέλος. Είναι οικονομική περισσότερο η ανάλυση αυτή και λιγότερο νομική. Αλλά θα συνεχίσουμε να κοιτούμε και τη διαφθορά από τη σκοπιά, τη νομική, ε, στο βαθμολόγιο που έχουμε, τον πίνακα επιδόσεων για τη δικαιοσύνη. Γιατί πρόσφατα προσθέθηκε ένα κεφάλαιο ε, για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν σε περιπτώσεις διαφθοράς στα κράτη-μέλη, πόσο καιρό χρειάζεται η απονομή της δικαιοσύνης. Άρα έχουμε αυτά τα δύο λοιπόν, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και τη δικαιοσύνη και το τρίτο θα είναι η ετήσια επισκόπηση. Και θα χρησιμοποιήσουμε διάφορες πηγές, όχι μόνο εκείνες που δίνουν τα κράτη-μέλη, τα στοιχεία, αλλά και από όλες πηγές αξιόπιστες, ε, τον Γκρέκο, ε, τον Όσα και τα λοιπά. Για το φορέα διοντολογίας, α, ήδη ξεπέρασα το χρόνο μου και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Ναι, ναι, τελειώστε. Απλώς ε, εγώ σας είπα ότι περάσετε το χρόνο σας. Αυτό... Ναι, αλλά το σφυράκι με αγχώνει λίγο. Ιδιαίτερα, γιατί θα ήθελα να μιλήσω τώρα για κάτι πολύ σπουδαίο. Ανεξάρτητο σώμα διοντολογίας χρειάζεται κάτι τέτοιο δεν ξέρω. Χρειάζεται μια τέτοια ομπρέλα ως φορέας. Ε, θα δω το δημοσιονομικό, μάλλον το κανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης, ε, ό,τι ισχύει ως προς τη δεοντολογία και θα δω τι θα ενταχθεί εκεί αν χρειάζεται ένα σώμα διοντολογίας. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και να προβαίνει στις συστάσεις για τα μέτρα που θα πρέπει να ε, λαμβάνονται ε, σε σχέση με κυρώσεις και ε, επιβολή τους. Αυτά ακόμα είναι σε εμβρυϊκό στάδιο. Πάντως είμαι ιδιαίτερα προσιλωμένη προς αυτή την προσπάθεια. Παρακαλώ, κύριε Φρόιντ, και θα αρχίσω το συντομότερο να εργάζομαι. Ο κύριος Φρόιντ. Ευχαριστώ. Συμπληρωματική ερώτηση για αυτά που είπατε προηγουμένως ε, σχετικά με το Μητρό των Λόμπι, το Μητρό διαφάνεια. Αυτό ήταν φιλοδοξία και της προηγούμενη Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι υποχρεωτικό αυτό το Μητρό των Λόμπι, αλλά και ε, στην περασμένη Επιτροπή ε, στις ε, επιστολές ανάθεση εντολή υπήρξε μια διατύπωση ε, ως προς την εξέβρεση μιας ισορροπίας απέναντι σε εκπροσώπους οικονομικών συμφερόντων. Στις νυν επιστολές ανάθεση εντολή έχει εξαφανιστεί αυτή η διατύπωση. Εσείς πώς το βλέπετε και ποιος είναι ο βασικός στόχος. Δεν είναι τελικά να μπει και το Συμβούλιο μέσα σε αυτό το πλαίσιο των Μητρών Διαφάνειας των Υποχρεωτικών. Εσείς κυρία Γιώροβα. Μάλιστα. Θέλω να μπει και το Συμβούλιο. Ε, τουλάχιστον να έρθει στη στρογγυλή τράπεζα και να το συζητήσουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν ίσοι κανόνες παιχνιδιού, οι ίδιοι για όλους. Διάβασα τις εκθέσεις, ε, μάλλον τα πρακτικά των συζητήσεων στο Συμβούλιο ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα και κατάλαβα ότι δεν θα είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Έχουν δίκιο και τα κράτη-μέλη. Ε, υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα στην πλήρη διαφάνεια αφενός και αφετέρου στη δυνατότητα να κάνεις διαπραγματεύσει με τρόπο αποτελεσματικό. Έχουν και αυτοί το δίκιο τους και το καταλαβαίνω. Είμαι απόλυτα έτοιμη να αρχίσουμε ένα τέτοιο διάλογο. Για την ισορροπία στην οποία αναφερθήκατε, δεν ξέρω γιατί έχει εξαφανιστεί αυτή η διατύπωση. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Σας ευχαριστώ. Στη συνέχεια, για ένα λεπτό, ο κύριος Νίκολας Φέστ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Γιώροβα. Είστε αρμόδια για τις αξίες και τη διαφάνεια, αλλά η ερώτησή μου είναι ως εξής. Πώς κατανοείτε εσείς τις αξίες ε, δηλαδή το πνεύμα των καιρών που και είναι μόδα αυτό τον καιρό και μπορεί να είναι ε, οτιδήποτε ε, έτσι ελαφρύ. Ε, είστε υπέρ και των συντηρητικών δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα του αγέννητου παιδιού. Κάτι τέτοιο θα ήθελε μια χριστιανική Ευρώπη. Ενώ οι αριστεροί μου φίλοι, οι σοσιαλιστές, οι φιλελεύθεροι και οι πράσινοι ε, ε, πράγματα ε, για τις ζωές των προσφύγων. Έχουν δικαίωμα στη ζωή όμως και τα γέννη τα παιδιά. Εσείς αυτά θα τα προσπίσετε. Ευχαριστώ. Απάντηση, κύριε Γιώροβα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φέστ. Ε, το δικαίωμα ε, το γέννη του παιδιού είναι στη δικαιοδοσία των κρατών μελών και την αρμοδιότητα. Αυτό ήτανε, μάλιστα. Παρακαλώ, έχετε ένα λεπτό, κύριε Φέστ, για συμπληρωματική ερώτηση. Κυρία Γιώροβα, εδώ και χρόνια διάφορα πράγματα τα θεωρήσατε φοβίες. Ομοφοβία, τρανσφοβία και διάφορες άλλες φοβίες και ιδιαίτερα Ισλαμοφοβία. Την περασμένη εβδομάδα στο Παρίσι ένας μουσουλμάνος σκότωσε τέσσερις αστυνομικούς και στο Βερολίνο επιτέθηκε ε, κάποιος ε, με ένα ε, στρατιωτικό μαχαίρι, πολεμικό μαχαίρι, δυνάμεις ασφαλείας μιας συναγωγής φωνάζοντας «Αλάχου Ακμπάρ». Ποια φοβία, είναι γεγονός αυτό. Και επίσης το Άρτε είχε ένα ρεπορτάζ που έδειχνε πώς το Κατάρ επηρεάζει την Ευρώπη με χρηματοδότηση για να εξισλαμιστεί. Τι λέτε λοιπόν για αυτές τις δολοφονίες, τα ε, φαινόμενα αυτά τα θεωρείτε ακόμα φοβίες ψυχοσικές ή μήπως έχει έρθει να καταλάβετε ότι είναι πραγματικότητα και να επιληφθείτε. Έχετε και εσείς ε, και πάλι το λόγο κυρία Γιώροβα. Ευχαριστώ και πάλι κύριε Φέστη για τη δεύτερη ερώτησή σας. Οι επιθέσεις και οι δολοφονίες είναι απολύτως απαράδεκτες. Ανεξαρτήτως ε, δράστη. Όταν γίνεται λόγος για ισλαμιστική τρομοκρατία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είδαμε να γίνονται πολλά για να προστατεύονται οι πολίτες από αυτούς τους τρομοκράτες. Και εγώ ήδη εργάζομαι και, και στα ψηφιακά γιατί και έχω τις στατιστικές ότι γύρω στο 20% των Ισλαμιστών ριζοσπαστικοποιούνται στη φυλακή και γύρω στο 80% στο διαδίκτυο. Κάναμε πολλά για να αυξήσουμε την κυβερνοασφάλεια και με την Europol και με τις αρμόδιες διεκτικές αρχές στα κράτη-μέλη. Πραγματικά κάνουμε πολλά για να μειωθεί ο κίνδυνος και το ρίσκο, αλλά θα πρέπει και πάλι να σας πω ότι όλες αυτές οι επιθέσεις και οι δολοφονίες είναι απαράδεκτες και θα πρέπει να εργαστούμε προς την αύξηση της ασφάλειας των Ευρωπαίων. Γιατί όταν ρωτάτε τους Ευρωπαίους τι περιμένουν από εμά, είναι ευημερία, ασφάλεια και σταθερότητα. Αυτό είναι το τρίπτυχο και αυτό είναι και η υποχρέωσή μας. Ευχαριστώ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Ασίτα Κανκό. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Γιώροβα, η παραπληροφόρηση είναι από τις πιο περίπλοκες προκλήσεις που έχει σήμερα αντιμετωπίσει η δημοκρατία μας. Σωστά το τονίσατε. Ε, τι αξίζει ακόμα η ελευθερία της έκφρασης όταν ο κόσμος δεν έχει τη σωστή πληροφόρηση. Αν θέλουμε μια ανοιχτή και ειλικρινή ε, συζήτηση και διάλογο που είναι απαραίτητη στην δημοκρατία θα πρέπει να προσέχουμε την παραπληροφόρηση αυτή γίνεται με τρόπο ύπουλο και είναι δύσκολο πολλές φορές να το ανακαλύψει, να το αισθανθεί αυτό και να δει που είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και το ψέμα. Οδηγεί σε σύγχυση τον κόσμο, τους κανονικούς πολίτες, τους δημοσιογράφους κτλ. Όλο και περισσότερες κυβερνήσεις, αν ζητάτε μάλλον από την κυβέρνηση, κυβερνήσεις και τις πλατφόρμες να είναι διαιτητές, δεν πρόκειται αυτό να βοηθήσει. Ε, θα πρέπει να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όσο περισσότερο εμπιστεύονται ε, την Ένωση οι πολίτες, τόσο καλύτερα θα καταπολεμούμε την παραπληροφόρηση. Εσείς πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα της εμπιστοσύνης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεδομένου και του ρόλου που έχετε για περισσότερη διαφάνεια. Έχετε το λόγο, κυρία Γιούροβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Κάνκο, για την ερώτησή σας. Ε, ήταν το θέμα και θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο σύντομη. Παραπληροφόρηση. Πώς ορίζουμε την παραπληροφόρηση για την οποία ε, κάτι πρέπει να κάνουμε πρέπει να μπορούμε να επαληθεύσουμε ότι είναι ψευδής ή παραπλανητική με στόχο πολιτικό, ε, πολιτική βλάβη να απειλήσει τη δημοκρατία, να υποσκάψει τις πολιτικές στην υγεία, το περιβάλλον και την ασφάλεια. Ε, αυτό είναι μια νέα απειλή και δεν θέλουμε όμως να την αντιμετωπίσουμε περιορίζοντας την ελευθερία έκφρασης και γι' αυτό έχουμε και πολύ ισχυρή στήριξη από τους πολίτες γιατί λένε διάφορες μελέτες ότι αυτό που θέλουν να κάνουν, θέλει ο κόσμος να κάνουμε για την παραπληροφόρηση είναι να εκπαιδεύσουμε καλύτερα τον κόσμο. Ακούγεται αλαζονικό αλλά εννοώ ότι πρέπει να επιτρέψουμε στον κόσμο να καταλάβει πότε χειραγωγείται, να τον εκπαιδεύσουμε ώστε να καταλαβαίνει πότε χειραγωγείται, να μπορεί να εντοπίσει την πηγή της πληροφορίας, να εντοπίσει ποιος είναι ο στόχος και οι προθέσεις. Δηλαδή να μπορεί να προσανατολιστεί καλύτερα στο ε, ψηφιακό κόσμο. Και αυτό οδηγεί στο να έχουμε μια πιο ε, ανθεκτική κοινωνία που θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους απειλές. Θέλουμε να εστιάσουμε στην παραπληροφόρηση ως νέα απειλή από δύο ε, πτυχές. Πρώτον, είναι η ένταση. Ένταση σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει, να υπάρχει παραπληροφόρηση που μπορεί να αποτελεί απειλή και για την ασφάλεια. Και εδώ θέλουμε να δουλέψουμε περισσότερο σε αυτή την ε, πτυχή πριν τις εκλογές ήμασταν έτοιμοι να αρχίσουμε να λειτουργούμε ένα τέτοιο σύστημα. Ε, δεν είχαμε τέτοια ε, προετοιμασία πριν τις ευρωεκλογέ, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι τώρα και πρέπει να συζητήσουμε την πτυχή της ασφάλειας και με τον ΝΑΤΟ. Έπειτα να δημιουργήσουμε την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και όσον αφορά την ε, χρονισμό, ειδικά πριν από τις εκλογές έχουμε περισσότερη παραπληροφόρηση και όλα είναι και περισσότερο τα πολιτικά κόμματα ε, είναι πολύ δραστήριοι παραγωγή ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης. Οπότε χρειάζεται να μπορούμε να αντιδράσουμε και θέλουμε να δούμε τους κανόνες για τις πολιτικές εκστρατείες και εδώ βλέπουμε πολύ συγκεκριμένα βήματα για να προχωρήσουμε. Κυρία Γιούροβα, σας θυμίζω να κοιτάτε και πόσο οπτητικός είναι ο χρόνος που έχετε για να απαντήσετε. Ε, περνά πολύ γρήγορα. Κυρία Κάνκο, πραγματικά καλό είναι που εστιάζεται στην προστασία των ανθρώπων και στην ευαισθητοποίηση των πολιτών. Αλλά αναρωτιέμαι, διαφάνεια θα σημαίνει θα είμαστε εκτεθειμένοι απέναντι σε hackers τι θα κάνετε ε, για να αντιμετωπίσετε με τους συναδέλφους σας ε, το ηλεκτρονικό έγκλημα. Επίσης, ε, στην οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο, τι ρόλο θα παίξουν οι πλατφόρμες και οι πάροχοι για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Δηλαδή, να κρατάνε και μικρό καλάθι οι πολίτες όταν βλέπουν κάτι στο ίντερνετ, να μην τα παίρνουν όλα τις μετρητής. Μάλιστα, σας ευχαριστώ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Θα πρέπει να σας πω ότι προσβλέπω στη συνεργασία με τη Μάργαρετ Φεστχάγκερ και την κυρία Γκουλάρα, διότι γιατί νομίζω πως θα ήταν πολύ θετικό να βρούμε τη σωστή ισορροπία για να καταλήξουμε σε ένα κοινό ορισμό για την ευθύνη των πλατφορμών. Η οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια πολύ ισχυρή νομοθεσία που λέει όμως ότι οι πλατφόρμες δεν είναι υπεύθυνε για το περιεχόμενο εκτός για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. Και αυτό εκεί είναι που πρέπει να το διευκρινίσουμε και να έχουμε μια ισχυρότερη νομοθετική όθηση ώστε να αυξηθεί η ευθύνη των πλατφόρμων. Εγώ είμαι πεπισμένη πως χρειάζεται ένα τέτοιο μέσο. Και την πρώτη ε, σκέλος, συγγνώμη αλλά δεν το κατάλαβα, δεν το θυμάμαι. Μικρόφωνο παρακαλώ, ναι. Πολύ συγκεκριμένα και σύντομα παρακαλώ. Ναι, αυτό προσπαθώ. Ναι, το πρώτο σκέλος ήταν το γεγονός ότι η διαφάνεια δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε γυμνοί όταν προσπαθούν να μας επιτεθούν οι hacker. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπιστεί η κυβερνοεγκληματικότητα και οι hacker. Όχι, είναι βεβαίως όχι και έχουμε... Ε, πρέπει να αυξήσουμε της, την τεχνική προστασία κατά του hacking σε όλα τα κράτη-μέλη. Οι επενδύσεις δεν αρκούν ακόμα, αλλά γίνονται κάποιες προσπάθειες, κάποια βήματα κατά του hacking. Και η αύξηση της ασφάλειας είναι στρατηγικά βήμα για όλα τα κράτη-μέλη Και δεύτερον, Τώρα, το να χρησιμοποιούμε το ψηφιακό χώρο είναι νομίζω πια ασφαλές γιατί έχουμε τον κανονισμό που προβλέπει πολύ ψηλές ε, ε, κυρώσεις και πρόστιμα. Νομίζω πως ε, από αυτή την άποψη οι Ευρωπαίοι είναι οι πιο ασφαλείς άνθρωποι στον πλανήτη. κυρία Στάτλερ, στα αγγλικά. Κύριε υποψήφια αντιπρόεδρε, ξέρετε ότι συνεργαστήκαμε στην Αυστριακή Προεδρία και συνεργαστήκαμε για πολλές αναταράξεις που είχαμε και ανησυχητικές εξελίξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία σε κάποια κράτη-μέλη. Ε, είπατε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δημοκρατία μας απειλείται. Μπορείτε λοιπόν να πείτε με ασφάλεια ότι η Επιτροπή σας θα ε, σταθεί στην Ευρώπη των αξιών και στον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής. Και να σας δώσω και ένα παράδειγμα για μια επίθεση ε, hacker που έγινε τον Αύγουστο του 2019. Συμφωνείτε λοιπόν ότι υπάρχει πιεστική ανάγκη να συντονίσουμε καλύτερα τις δυνάμεις μας και την ενέργειά μας για να προστατεύσουμε τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα και να αυξήσουμε τη συνεργασία μεταξύ κρατών μαλλών. Και εν και ερώτησης ε, συμπληρωματική στην προηγούμενη ερώτηση, θεωρείτε ότι πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να υπάρχει ταχύ αντίδραση σε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα όταν έχουμε επίθεση κατακρίσιμων υποδομών. Δύο λεπτά για να απαντήσετε, κυρία Γιούροβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κυρία Στάτλερ. Πρέπει να πω ότι έχουν γίνει πολλά για να προστατεύσουμε τα δίκτυά μας και τον κυβερνοχώρο μας ε, κατά του hacking και θα πρέπει να γίνουν και άλλα ακόμα. Υπάρχει αρχιτεκτονική δομή, ο ΕΝΗΣΑ συντονίζει τις δράσεις ε, των κρατών μελών που ε, έχουν φορείς που επικεντρώνονται στην κυβερνοασφάλεια. Θεωρώ ότι η συνεργασία λειτουργεί πολύ καλά, αλλά όπως σας είπα και προηγουμένως υπάρχουν και ανάγκη για πολύ περισσότερες δυνατότητες στα περισσότερα κράτη-μέλη. Το γεγονός ότι υποτιμούμε το θέμα αυτό ε, πάντα τιμωρείται πολύ αυστηρά από τις συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες αναφέρατε. Και έχουμε συγκεκριμένη νομοθεσία που θα πρέπει να αναθεωρηθεί το 2021. Έχουμε την οδηγία η οποία προστατεύει τις κρίσιμες ουσιαστικές υποδομές ε, και αναφερθήκατε και στη συγκεκριμένη υπόθεση το γεγονό ότι ε, τα πολιτικά κόμματα δεν προστατεύονται από τη συγκεκριμένη οδηγία. Σω αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη στην αναθεώρηση συγκεκριμένη οδηγία. Ωραία, ευχαριστώ. Κύριε Ετστάτλερ, το δεύτερο λεπτό σας. Υπάρχει και αύξηση του αντισημιτισμού που αποτελεί απειλή για τι κοινέ μας αξίες ε, και για την κοινωνία μας συνολικά. Ε, ευπρόσδεκτα τα μέτρα τα οποία λήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατεπολέμηση του αντισημιτισμού και το γεγονό ότι θα πρέπει να υπάρχει και συντονιστή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ορίστηκε και ήταν κομβικό ο ρόλο τη ε, που οδήγησαν και στι ε, δηλώσει του Συμβουλίου για την καταπολέμηση αντισημιτισμού το Δεκέμβριο του 2018. Αυτή η δήλωση τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση ασφαλεία και για πρώτη φορά να φέρει έναν γενικό δεσμευτικό ορισμό του αντισημιτισμού. Υπάρχουν πάρα πολλέ προκλήσεις ακόμα, κυρίως ότι πρέπει να ε, δια ασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει και ασφάλεια σε αυτή την περίπτωση. Σκοπεύετε να ενισχύσετε και να αναβαθμίσετε την εντολή αυτού του συντονιστή ε, για την ε, νέα θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τι περαιτέρω βήματα σκοπεύετε να αναλάβετε. Κύριε Γιούροβα, ευχαριστώ πολύ. Να σας πω ότι ο αντισημιτισμός δεν είναι ένα θέμα στο οποίο μπορώ να επεκταθώ μέσα σε ένα λεπτό. Θα προσπαθήσω. Είναι πονήριστη αυτή η ιστορία για την Ευρώπη. Οι Εβραίοι πολίτε ε, φεύγουν και πάλι από την Ευρώπη γιατί φοβούνται. Και υπάρχει και μια έρευνα στην οποία διαπιστώνουμε ότι το 80% των Εβραίων που διαμένουν στην Ευρώπη έχουν ε, σοβαρό πρόβλημα. Και το πιο πιεστικό ζήτημα είναι η ασφάλειά τους αν ρωτήσετε άλλους Ευρωπαίους θα σας πούνε ότι είναι πραγματικά ε, η υγεία, η θέση εργασίας για τους Εβραίους είναι η ασφάλειά τους. Γι' αυτό λοιπόν λαμβάνονται πολλά μέτρα. Υπήρχε και ο ορισμός του συντονιστή, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το Δεκέμβριο πέρσι οι Υπουργοί Εσωτερικών και Εσωτερικών Υποθέσεων δεσμεύτηκαν μέσω μιας δήλωσης ότι θα υπάρξουν εθνικές στρατηγικές για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Συζητήσαμε θέματα ασφαλείας σε μια ομάδα εργασίας φέστος με τους υπουργούς και τους αρμόδιους εταίρους διότι υπήρξε δέσμευση από τους ίδιους τους υπουργού για αύξηση του προπολογισμού για προστασία ε, χώρων στους οποίους συχνάζουν Εβραίοι, συναγωγές, τα σχολεία τους κλπ. Αλλά ε, πρέπει να γίνουν ακόμα κι άλλα. Έχουν γίνει πολλά, ο αντισημιτισμός αυξάνεται και φυσικά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να είμαστε απόλυτα σαφείς και να στέλνουμε ένα μήνυμα ότι είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Ωραία, σας ευχαριστώ και τώρα περνάμε Στη, Ραμό, στη Ραμόνα Στρουγκάριου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επίτροπε Γιούρεβα. Ελευθεροτυπία, πλουραλισμό και ελευθερία έκφραση είναι, είναι θεμέλια κάθε δημοκρατία. Και ωστόσο είναι υποεπίθεση εδώ και τώρα, εδώ στην Ευρώπη. Την ώρα που μιλάμε, η ερευνητική δημοσιογραφία στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει τεράστιε πιέσει στη Βουλγαρία λόγω των ε, ερευνών τους και καθώ ε, μιλάμε ο χώρος για την ελευθερία έκφραση ε, περιορίζεται στι χώρες μα, συρρυκνούται. Ποια μέτρα θα αναλάβετε ώστε να εμποδίσετε επιθέσεις κατά δημοσιογράφων και να εξασφαλίσετε την ασφάλειά τους. Θα προτείνετε μια πανευρωπαϊκή νομοθεσία, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε και θα δεσμευτείτε για ένα μόνιμο ταμείο για την ερευνητική δημοσιογραφία και την ελευθεροτυπία εντός του πρώτου έτους της θητείας σας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Στρουγκάριο. Στην πρώτη ο έτος της εντολής μου θα εργαστώ εντατικά για το σωστό σχεδιασμό του προγράμματος χρηματοδότησης υπό το πρόγραμμα Creative Europe, Δημιουργική Ευρώπη, που στόχο έχει να στηρίξει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Προβλέπονται 61 εκατομμύρια για 7 χρόνια. Οπότε πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσο γίνεται πιο αποδοτικά τα χρήματα αυτά, ώστε να έχουμε συστημικά και συστηματικά μέτρα που θα καλύψουν όλα τα κρατημέλη και θα προστατέψουν καλύτερα του δημοσιογράφου σε περιπτώσεις όπου τα συστήματα τα κρατικά μπορεί να θέτουν σε κίνδυνο τη, δημοσιογραφία, αλλά και με μονομένες απειλές προς μεμονωμένους ε, ε, δημοσιογράφους. Ε, θα εργαστούμε λοιπόν για αυτό το είδος την χρηματοδότηση και θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε μια σωστή χαρτογράφηση, γιατί υπάρχουν πολλές μεταβλητές Θα εξετάσουμε τη δυνατότητα ε, εξυγχρονισμού της νομοθεσίας. Διαβλέπουμε δυνατότητες στο διεθνές ε, ε, δίκαιο αλλά θα εξετάσουμε και τη δυνατότητα για δημιουργία ενός συστήματος νομικής αρρωγής ή μιας γραμμής βοήθειας για δημοσιογράφους που, είναι, που απειλούνται, γιατί η κατάσταση είναι πολύ ανησυχητική. Καθημερινά παίρνω ε, mail από τις ενώσεις δημοσιογράφων και ακούω φρικτές ιστορίες. Καταρχάς ε, κοιτάω να δω αν είναι από την Ευρώπη ή συνήθως προέρχονται εκτός Ευρώπης αλλά και από την στην Ευρώπη και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Βεβαίως τα μέσα, ο πλουραλισμός και η παρακολούθηση θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Θα έχουμε άλλη μια εντολή για το 2020, θα έχουμε καλύτερη χαρτογράφηση για το τι συμβαίνει στα κατημέλη και ίσως και έμπνευση για το τι μπορούμε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρία Σρουγκάριου, έχετε και πάλι το λόγο για επερώτηση. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Η απάντησή μου σχετίζεται με την ε, επερώτησή μου, γιατί ξέρετε ότι σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις οι απειλές και ο εκφοβισμός δημοσιογράφων προέρχεται από τους, τα ίδια τα, ε, τους, τους ίδιους τους ερευνόμενους και από τις εθνικές αρχές. Πώς μπορεί να προστατευτούν οι δημοσιογράφοι εφόσον δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις εθνικές αρχές. Μήπως είναι καιρός να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. Κατάλαβα, δεν κατάλαβα λέει η Επίτροπος, οι απειλές από που προέρχονται απειλούνται αλλά δεν μπορούν να βασιστούν στις εθνικές αρχές. Μπορεί δηλαδή η απειλή να προέρχεται από τι ίδιε εθνικέ αρχέ τι οποίε ερευνούν. Πολύ δύσκολη η ερώτησή σα αυτή και δεν θα παραστήσω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξοπλιστεί με ισχυρές ε, νομοθετικές ή εκτελεστικές εξουσίες σε αυτές τις περιπτώσεις, για τέτοιες μάλλον περιπτώσεις. Πολύ με ανησυχεί όταν ακούω κάποιους ε, πολιτικούς ε, που επιτίθενται προφορικά σε δημοσιογράφους διότι δεν τους αρέσουν αυτά που γράφουν οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι Ε, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται σε τέτοια θέση. Όταν να σε κάποια κράτη-μέλη ε, ε, δέχονται προφορικές επιθέσεις και επιγραμμικά, είναι απαράδεκτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει επαρκείς αρμοδιότητες για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά όπως είπα πριν θα εξετάσω τη δυνατότητα πιο αποτελεσματικής χρηματοδότησης ώστε να βοηθηθούν αυτοί που το χρειάζονται και οι, οι δημοσιογράφοι που απειλούνται με συστηματικό και μεθοδικό τρόπο. Υπήρξε μια ενδιαφέρουσα έρευνα ε, από τη διάσκεψη ερευνητικής δημοσιογραφίας που έγινε πρόσφατα στο Αμβούργο και εκείνοι είπαν τα εξή ότι χρειάζεται περισσότερη διασυνοριακή συνεργασία ανάμεσα στους δημοσιογράφους και τις ενώσεις τους και θα πρέπει να υπάρξει και περισσότερη αλληλεγγύη μεταξύ των ίδιων των δημοσιογράφων. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε εμείς να εγγυηθούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σίγουρα είναι ένας τρόπος για να προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ο, ο κύριος Λέβε έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακούω συνεχώς ότι η βασικότερη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι βασίζεται σε κανόνες αυτός ο οργανισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα, έχει δεσμευθεί να σέβεται τις αρχές του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ είναι ξεκάθαρα. Κανένα κράτος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει οικονομική, πολιτική ή άλλη ε, ε, ισχύει για να επιβάλλει σε κάποιο κράτος μέλος διάφορα πράγματα. Ε, έχετε ε, απορρίψει την πρόταση του Μπόρις και ε, πραγματικά δεν ε, ε, επιβάλλεται απλώς την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μεγάλη Βρετανία, μιλώντας για το backstop της Ιρλανδίας, ότι θα πρέπει να συμφωνήσει η τοπική κυβέρνηση το Stormont. Η Βόρεια Ιρλανδία είναι το πτήμημα που θα πρέπει να πληρώσουμε εμείς για να φύγουμε από αυτή τη λέσχη. Για να απαντήσει η Επίτροπος έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Λεβε για τις ερωτήσεις σας. Θα απαντήσω ως εξής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, ε, κάτι, ε, μια ένωση όπου οι αξίες έχουν πάντα νόημα. Ε, πάντα δρούμε με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο, το πρωτογενές και το δευτερογενές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι θεματοφύλακα των συνθήκων. Αυτές είναι οι αρχές που χρησιμοποιούμε και σε όλες τις διαπραγματεύσεις για το Brexit που είναι πάρα πολύ δύσκολες και τώρα βρίσκονται ε, σε μια ε, φάση πάρα πολύ ε, δύσκολη. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πραγματικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πάντα υπερισχύουν οι αξίες και οι αρχές και ποτέ δεν θυμάμαι κατάχρηση των αξιών ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης εις βάρος κάποιου κράτους μέλους ή ως τιμωρία, όπως το αναφέρετε. Διαφωνώ βαθύτατα με τα όσα είπατε. Ευχαριστώ. Ερώτηση κύριε Λεωβέ, συμπληρωματική. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε, αλλά πολύ καινότοπα. πώς ε, ορίζονται οι αρχές και πώς κρίνονται με βάση αυτά που λέμε ή αυτά που κάνουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβεται απολύτως το διεθνές δίκαιο. Ε, να το συγκεκριμενοποιήσω. Με βάση το διεθνές δίκαιο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει δικαίωμα να αλλιεύει μετά το Brexit στα ε, χωρικά μας ύδατα εκτός αν υπάρξει συμφωνία. Και είτε υπάρχει είτε όχι συμφωνία δεν μπορεί να γίνεται διάκριση μεταξύ των μελών του ΠΟΕ. Τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν υπάρξει συμφωνία να ισχύει το διεθνές δίκαιο έτσι ώστε να μην μας κλέβουν οι Ολλανδοί ψαράδες τα ψάρια μας από τα χωρικά μας ύδατα και οι Γάλλοι ε, ε αλληλείς να μην μπλοκάρουν ε, το καλέ. Ε, απάντηση. Thank you very much for your Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Θα παραπέμψω την ερώτηση αυτή στον συνάδελφό μου Σελ Μπαρνιέ που είναι διαπραγματευτής και γνωρίζει όλα τα θέματα της συμφωνίας, της μη συμφωνίας, της όποιας συμφωνίας. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, η κυρία Γιόντσεβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πρόσφατα οι μάρτυρες δημοσίου συμφέροντας αποτέλεσαν σημαντική πηγή ε, πληροφοριών, τα LuxLeaks, τα Panama Papers, ε, το Cambridge Analytica κλπ. Αυτοί λοιπόν οι μάρτυρες ε, ανακάλυψαν παράνομες πρακτικές όπως η προστασία δεδομένων, η διαφθορά, φοροδιαφυγή, έλλειψη προστασίας, ασφάλεια τροφίμων, δημόσια υγεία και τα ανέφεραν αυτά τα γεγονότα. Η πρόσφατη οδηγία για την προστασία των μαρτύρων δημοσίου συμφέροντο του επιτρέπει να μιλήσουν άμεσα με τον τύπο ε, υπό συγκεκριμένε προποθέσει. Τι κατευθυντήριες γραμμέ θα δώσετε προ τα κράτη-μέλη όσον αφορά την οδηγία και την εφαρμογή τη. Πώ θα εξασφαλίσουμε ότι κατά την εφαρμογή τα κράτη-μέλη δεν θα υπεβάλλουν ε, υπερβολικά περιοριστικέ διαδικασίε ε, που ουσιαστικά θα κάνουν αδύνατη την δημόσια αποκάλυψη πληροφοριών για του μάρτυρε δημοσίου συμφέροντο. Πώ θα εξασφαλίσετε την ελευθερία της έκφρασης για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Ευχαριστώ. Έχετε το λόγο, κυρία υποψήφια επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Δυστυχώς δεν άκουσα σήμερα τη συζήτηση στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης. Φαντάζομαι ότι θα έγινε μια συζήτηση γιατί η οδηγία ε, εγκρίθηκε μετά από τις διαπραγματεύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να φρεσκάρω λίγο τις γνώσεις μου για το πώ προετοιμάζονται τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας ε, ε, στο εθνικό του σύστημα. Αλλά προβλέπω ότι θα τη λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη διότι η οδηγία αυτή επιβάλλει πολύ συγκεκριμένε υποχρεώσει προ τα κράτη-μέλη και προ τα θεσμικά όργανα. Υπάρχει υποχρέωση, για παράδειγμα, να ανοίξει ο εσωτερικό δίαβλο που θα πρέπει να είναι ο πιο εγγύς στο μάτρα δημοσίου συμφέροντο, ο οποίο θέλει να καταγγείλει κάποια ε, παρανομία στο χώρο εργασία. Δεν αφορά αυτό του δημοσιογράφου αλλά ανθρώπου οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με κάτι στραβό στο χώρο τη εργασία του και θέλουν κάπου να το ανακοινώσουν. Πρόκειται για θαραλέου ανθρώπου που αξίζουν προστασία Γι' αυτό ακριβώ ε, και προετοιμάσαμε πάρα πολύ προσεκτικά πρώτα τον εσωτερικό διάβλο εντός του θεσμικού οργάνου. Μετά, εάν αυτός δεν είναι αξιόπιστος ή ασφαλός, ε, ή ασφαλής ή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τους εξωτερικούς διάβλους, οι οποίοι θα πρέπει ε, να είναι αυτοί που θα προετοιμάσουν τα κράτη-μέλη. Αυτή είναι η υποχρέωση του κράτους να ετοιμάσει ένα διάφανο, ασφαλή διάβλο για να αποκτήσουν πληροφορίες από τους μάρτυρες και ε, ως ίστατη καταφυγή να προσφύγουν στα μέσα ενημέρωσης. Νομίζω ότι αυτό το σύστημα θα αυξήσει δραστικά την προστασία αυτών των θαραλέων ανθρώπων, αυτών των μαρτύρων, οι οποίοι δεν μπορούν να ασιοποιήσουν όταν συμβαίνει κάτι φρικτό, ένα έγκλημα κατά του περιβάλλοντος, όταν υπάρχει φοροδιαφυγή ή κάτι αντίστοιχο. Είχα το προνόμιο να συναντηθώ με κάποιους από τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος ε, σε μεγάλες υποθέσει και θαυμάζω το θάρρος τους και πιστεύω ότι ε, τους χρειάζεται πραγματικά πολύ καλύτερη προστασία. Πιστεύω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη θα κάνουν ό,τι μπορούν εγκαίρω. Για δεύτερο λεπτό έχετε το λόγο. δημοσιογράφοι, ε, απλοί πολίτες, ε, πολιτικοί, ακτιβιστές μπορεί να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος. Πώς θα εξασφαλίσετε ότι η νομοθεσία θα προστατεύει τους πάντες αποτελεσματικά. Θα εσμεύεστε να προωθήσετε προγράμματα που θα παρέχουν χρηματοοικονομική βοήθεια σε αυτούς που μπορεί να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, ε, νομικές ε, διαδικασίες και να πρέπει να πληρώσουν ε, τα νομικά έξοδα όταν ε, κάνουν τη δουλειά τους. Θα εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά πώς θα σχεδιάσουμε το τμήμα του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη που αφορά την προστασία της ανεξάρτητης δημοσιογραφίας ε, και το πρόγραμμα για τις αξίες και την ηθαγένεια που προστατεύει την ε, ε, ενεργό κοινωνία των πολιτών. Ο τρόπος με τον οποίο θα σχεδιάσουμε τα προγράμματα θα είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγων για την αποτελεσματικότητα της χρήσης αυτών των κονδυλίων. Και εγώ θέλω τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιηθούν για πράγματα που χρειαζόμαστε. Αν χρειαζόμαστε περισσότερη προστασία για τους δημοσιογράφους και για τους ανθρώπους που απειλούνται από διάφορους κύκλους ε, και από κάποιους που δεν θα τους χαρακτήριζα αντιπάλους, αλλά ανθρώπους που τους απειλούν για παράδειγμα στο διαδίκτυο, θα πρέπει να σκεφτούμε με έξυπνο τρόπο πώς μπορούμε να παρέχουμε νομική συνδρομή, αλλά και ε, προστασία, φυσική προστασία και φυσικά αυτό θα μπορούσε να γίνει και με ευρωπαϊκά χρήμα. Και εγώ θα συζητήσω με τα κράτη-μέλη για μια πρόταση συγχρηματοδότησης, διότι αυτό δεν είναι θέμα μόνο Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να είναι και πολύ ισχυρή υποχρέωση για τα κράτη-μέλη. Πρέπει να προστατεύονται οι δημοσιογράφοι καλύτερα. Ελπίζω λοιπόν να έχει αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Μίλτσικ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Υποψήφια Αντιπρόεδρε, ήδη ακούσαμε την τελευταία έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που δείχνει ότι ο κόσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος ε, από τον τρόπο με τον οποίο εμείς καταπολεμούμε την παραπληροφόρηση στα ευρωπαϊκά μίντια. Συμφωνείτε πιστεύω όλοι ότι αυτό το θέμα της παραπληροφόρησης δεν είναι μόνο πρόβλημα για την ασφάλεια της ενημέρωσης αλλά και για την ίδια τη δημοκρατία μας. Θα συμφωνήσετε μαζί μου λοιπόν ότι δεν χρειαζόμαστε μεγάλα εργαλεία στις προεκλογικές περιόδους για να ε, καταπολεμούμε σε ευρία κλίμακα την παραπληροφόρηση, αλλά συγκεκριμένα μέτρα και μέσα στοχευμένα για να ε, αυξηθεί η ανθεκτικότητα της κοινωνίας και ε, οι δεξιότητες των πολιτών ως προς τα ψηφιακά. Ποια είναι τα συγκεκριμένα μέτρα λοιπόν που προτείνεται για να προστατεύετε τους δημοσιογράφους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχουμε στοχευμένες όπω όπως των δύο δημοσιογράφων στη Μάλτα και τη Σλοβακία και πώς τέτοια φαινόμενα μπορούν να αποφεύγονται και τι νομικές πτυχές ερωτώ και τι πρακτικές. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω από το τελευταίο. Πέρα από όλα αυτά που ανέφερα προηγουμένως, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη ε, χρηματοδότηση αυτή για συστηματική προστασία μαζί με τα κρατημέλη και υποστήριξη και φύλαξη των δημοσιογράφων. Θα ήθελα επίσης να ενθαρρύνω τους ίδιους τους δημοσιογράφους να ε, αναζητούν βοήθεια. Όταν υπάρχουν τέτοιες φρικτές απειλές εις βάρος και τα βία μέσα ε, ε, και τα απειλητικά μηνύματα που τους στέλνουν στο διαδικτύο, να μην διστάζουν, να απευθύνονται στην αστυνομία για να τα έρευνα αυτά τα φαινόμενα. Όταν κάποιος εκτοξεύει απειλές με τέτοιο τρόπο και με τέτοια ένταση, αυτό αφορά την ίδια τη βασική λειτουργία του κράτους που είναι η παροχή προστασίας προς τους πολίτες. Δηλαδή και αυτό θα είναι στοιχείο της δικής μου ε, στράτευσης, να συζητήσω με ενώσεις που ασχολούνται με αυτά τα θέματα, ε, ενώσεις δημοσιογράφων για να χρησιμοποιούν καλύτερα την προστασία είναι ευθύνη του κράτους να την εγγυάται. Υπάρχει λοιπόν δυνατότητα και για την πρώτη σας ερώτηση, πραγματικά, ε, δεν θα πρέπει να είμαστε ιστερικοί με αυτά τα θέματα της παραπληροφόρησης. Έχουμε τις πλατφόρμες ε, που έχουν τώρα ένα κώδικα ε, πρακτικής. μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου την άλλη εβδομάδα θα μου έχουν δώσει τα πρώτα στοιχεία πλατφόρμες για το τι συνέβη προεκλογικά πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές. Ε, θα αναλύσουμε τα αποτελέσματα και του χρόνου θα έρθουμε με μία πρόταση για να αυξηθεί και να αναβαθμιστεί το πρόγραμμα ε, δράσης για την παραπληροφόρηση. Αλλιώς θα συνεχίσουμε όπως ε, εργαζόμαστε αυτόν τον καιρό. Αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι απλώς επιβάλλοντας μια ε, υποχρέωση ε, στις πλατφόρμες θα λύσει τα προβλήματα. Αυτό είναι αφέλεια. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Θα πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμες λύσεις, ο κόσμος να μαθαίνει τις ψηφιακές δεξιότητες και τα μίντια και ε, αρχίσαμε με τους νέους και με τους ηλικιωμένους πρέπει να σας πω σε πολλές χώρες γιατί φοβούνται ε, και είναι και στόχοι. Αυτά είναι τα πιο μακροπρόθεσμα μέτρα που θα πρέπει να σκεφτούμε. Ε, Συμπραγματική ερώτηση ο κύριος Μπίλτσικ ε, Ευχαριστώ κυρία υποψήφια Αντιπρόεδρε. Στα Σλοβακικά τώρα μια συμπληρωματική ερώτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην τωρινή σας ε, θητεία ε, και στην ανεξαρτησία σας απέναντι στα κράτη-μέλη. Αυτή η ανεξαρτησία θα είναι πιο σημαντική τώρα, στη νέα σας θέση, που θα έχετε το χαρτοφυλάκιο της διαφάνειας και των αξιών, εάν επιβεβαιωθείτε, εάν εγκριθείτε. Το κράτος δικαίου λοιπόν, εάν απειλείται σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, είστε πολύ στεναροί από, απέναντι. Αυτό θέλω να ακούσω τουλάχιστον από εσά. Εξ όσων διάβασα, ε, με χαρά ε, στις γραπτές σας απαντήσεις, είστε διατεθειμένοι να συνεργαστείτε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ερωτώ, θα απορρίπτατε ε, τις απόψεις του Πρωθυπουργού της Τσεχικής ε, Δημοκρατίας ότι στο Κοινοβούλιο ε, γίνονται διάφορες ανόητες συζητήσεις όπως και στο Τσεχικό Κοινοβούλιο. Κατανοώ πάρα πολύ καλά αυτά που λέτε. Ε, γιατί κατανοώ τη Σλοβακική, γιατί οι άνθρωποι της ηλικίας μου καταλαβαίνουν Σλοβακικά. Ε, δύο απαντήσεις. Βεβαίως θα συνεχίσω ανεξάρτητα να ασκώ τα καθήκοντά μου. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Όχι μόνο στην περίπτωση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου των αξιών και του κράτους δικαίου. Ε, δεσμεύομαι ε, ότι θα συνεχίσω να το κάνω, απολύτως. Σε ό,τι αφορά τη γνώμη ότι τα κοινοβούλια είναι κάποιοι χώροι ο ματέων συζητήσεων, για να το πω λίγο πιο κομψά και κατεφημισμών, ε, βεβαίως και διαφωνώ βαθύτατα, είτε πρόκειται για τα Εθνικά Κοινοβούλια, είτε για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κοινοβούλια είναι απαραίτητο στοιχείο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, όπως και οι συζητήσεις που γίνονται. Ευχαριστώ. Και τώρα προχωρούμε. Επόμενη Ομιλήτρια η κυρία Κλέρ Ντέιλι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς, ε, όσοι πιστεύουν στο ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι, έχουν καθήκον να υπερασπιστούν τη συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής, ώστε οι Ιρλανδοί και από τις δύο πλευρές των συνόρων να συνεχίσουμε να ζούμε εν ειρήνη. Πάντως υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στους πολίτες της Ευρώπης και τους θεσμούς και ένας τρόπος για να γίνει αυτό θα είναι η ηθική και δεν ικανοποιήθηκα στην απάντηση, από την απάντησή σας για την ανάγκη δημιουργίας ενός ανεξάρτητου σώματος σώματος ηθικής. Πιστεύουμε πως είναι πολύ σημαντικό αυτό ε, και θεμελιώδες. Εσείς είπατε κάτι ότι θα είναι συμβουλευτικό σώμα και τα λοιπά, ενώ στη γραπτή σας ε, απάντηση είπατε ότι θα θεωρήσετε ότι η διοντολογία θα είναι μια ηθική υποχρέωση. Εσείς δεσμεύεστε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο ανεξάρτητο σώμα διοντολογίας. Πιστεύω πως είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη θητεία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντέιλι για την ερώτησή σας. Μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι ήθελα να πω για το ανεξάρτητο σώμα ε, ηθικής και διοντολογίας. Δεν είχα το χρόνο να τα πω όλα αυτά. Είπα πως ίσως να είναι μια από τις επιλογές ένα συμβουλευτικό σώμα το οποίο θα συστηθεί από ανεξάρτητους ε, ανθρώπους ε, με αξιοπιστία, ε, ανθρώπους εκτός των θεσμών που θα εξετάζουν με συγκεκριμένη βάση με γρήγορο τρόπο γιατί και εκεί έχει νόημα η ταχύτητα και γιατί πολλές φορές χρειάζεται λοιπόν μια γρήγορη αντίδραση των θεσμών. Το ανέφερα αυτό ως μία από τις πιθανές επιλογές. Η άλλη επιλογή όντας ότι οι θεσμοί θα συμφωνήσουν για ένα σώμα δεοντολογίας με ισχυρότερε αρμοδιότητες. Αλλά για να είμαι ειλικρινής, διάβασα κάποιες περιμένεις περιπτώσεις όπου δημιουργήθηκαν τέτοια σώματα και δεν υπήρχε ποτέ ισχυρή ε, στήριξη από τους θεσμούς. Δεν υπήρχε ανάγκη γιατί είχαν ε, το δικό τους εσωτερικό κανονισμό κάθε φορά δεν θέλω λοιπόν να προβλέψω οτιδήποτε εδώ, είναι κάτι το νέο. Θέλω να ξεκινήσω το διάλογο με τους θεσμούς, να εξετάσω τις παλιότερες προτάσεις και να βρούμε το καλύτερο δυνατό μοντέλο για έναν εξάρτητο σώμα διοντολογίας, το οποίο θα είναι όμως πολύ ισχυρό Θέλουμε να είναι ένας ισχυρός φορέας, ένας ισχυρό θεσμός που θα συνδημιουργήσει μαζί μας την ευρωπαϊκή πολιτική κουλτούρα. Γιατί πρόκειται και περί αυτού. Δεν θέλω να κλείσω καμιά πόρτα, απλά θέλω να πω θα το εξετάσουμε από κοινού, γιατί βέβαια δεν θα είναι μόνο δουλειά της Κομισιόν, θα είναι ένα από τα θέματα όπου μας περιμένει εντατικός διαθεσμικός διάλογος. Ευχαριστώ. Κυρία Ντέιλι, προταση. Ένα λεπτό. Αυτό που λέτε είναι ότι είστε δεσμευμένοι για ένα τέτοιο σώμα, αλλά δεν είστε βεβαία για το τι μορφή θα πάρει. Ελπίζω αυτό να εννοούσατε. Δεύτερη μου ερώτηση. Το, στο χαρτοφυλάκι σα έχετε την ευθύνη να υπερασπιστείτε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία από εξωτερική επέμβαση, αλλά και για τη στήριξη ανεξαρτήτων δημοσιογράφων. Ε, ξέρουμε ότι υπάρχουν ισχυρέ προστασίε στην Ευρώπη που μπορούν όμω να υποβαθμιστούν εάν ξένε δυνάμει επηρεάσουν εκτό Ευρώπη ε, ξέρουμε, ας πούμε, ότι το 2010 η Not for Profit δημοσίευσε, η Wikileaks έδωσε σπουδαία βραβεία για την ερευνητική δημοσιογραφία στη διάρκεια των πολέμων του Αφγανιστάν και του Ιράκ και τώρα ο εκπρόσωπο του Wikileaks είναι στη φυλακή στη Βρετανία και αντιμετωπίζει έκδοση στη ΣΥΠΑ που στόχο έχει να, ε, να ποινικοποιήσει τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής. Εσείς τι θα κάνετε για να στηρίξετε την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και την κοινωνία των πολιτών και την ελευθερωτική στερεοτυπία από ξένου μέρη όπως είπα, και ιδιαίτερα για να προστατεύσετε τους, ε, τους δημοσιογράφους εντός Ευρώπης από πολιτικές διώξεις. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό έχετε κυρία Γιούροβα. Φοβούμαι πως η έκδοση είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Εγώ δεν μπορώ να μπω σε εθνικά χωρικά ύδατα. Αναφέρομαι στην υπόθεση του κυρίου για ενώ αναμένουμε την απόφαση των του Βρετανικού Δικαστηρίου. Βεβαίως η Κομισιόν οφείλει να ε, γνωρίζει ποια είναι τα όρια των αρμοδιοτήτων της. Όσον αφορά την προστασία κατά καταχρηστικής ε, ε, σύγκρουσης ε, πρέπει να δούμε τις συγκεκριμένες υποθέσεις κάθε φορά ίσως να πρέπει να αναλύσουμε τις περιπτώσεις όπου οι δημοσιογράφοι έχουν να αντιμετωπίσουν πολύ δυσάρεστες διαδικασίες εκτός της Ένωσης αλλά πρέπει να δω και να χαρτογραφήσω αυτήν την, την κατάσταση πρέπει να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες Πρόεδρος Ωραία. Περνάμε τώρα στη Σίλβια Σπούρεκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύρια υποψήφια Πρόεδρε. οι ευρωπαϊκές συνθήκες ε, εξασφαλίζουν ε, διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την κοινωνία των πολιτών. Εσείς ε, έχετε αναλάβει το διάλογο με τις εκκλησίες και φιλοσοφικούς ε, και θρησκευτικού οργανισμούς ε, βάσει της επιστολής σας. Αλλά σε αυτή την επιστολή μόνο ο διάλογος με τις εκκλησίες ε, είναι τονισμένος με μαύρα γράμματα. Υπάρχει κάποια διάκριση ενώπιον των φιλοσοφικών και μη θρησκευτικών οργανώσεων. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τώρα έχει παραδεχτεί ότι υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες παρά το γεγονός ότι ήταν κατά των ε, γυναικείων, των ευρωπαϊκών αξιών, ε, των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ και των δικαιωμάτων των γυναικών. Τι θα κάνετε λοιπόν ώστε να εξασφαλίσονται ότι θα απορρίπτονται τέτοιες πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Κύριε Γιούροβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σπούρεκ. Ε, καταρχάς νομίζω ότι εμένα μου έχει ανατεθεί ο διάλογος με τις εκκλησίες και φιλοσοφικές ε, μη θρησκευτικέ ομάδες επίσης. Δεν υπάρχει λοιπόν κάποια προτίμηση προς τις εκκλησίες, ούτε προνομιακή μεταχείριση. Αυτό θα είναι ένας νέος κλάδος για μένα εν, εν μέρη. Εν μέρη διότι ε, έχω ουσιαστική εμπειρία από την προηγούμενη θητεία μου, ε, νομίζω η πρώτη το 2016, αν δεν κάνω λάθος, όπου είχαμε μία συζήτηση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και ε, καλέσαμε εκπροσώπους όλων των εκκλησιών. Και ήδη η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ενθαρρυντική. Μας απέδειξαν ότι μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους και μπορούν να συμφωνήσουν για τη σωστή άγουσα για θέματα αξιών. Επομένως ε, ήταν ιδιαίτερα σημαντικό και χρήσιμο όλο αυτό και όλη αυτή η εκδήλωση. Και επίσης, όταν προωθούσα την ε, σύμβαση της Κωνσταντινούπολης στα κράτη-μέλη, γιατί ασχολούμουν με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη σύμβαση της ε, Κωνσταντινούπολης και ήθελα να παρουσιάσω και τη σύμβαση στα κράτη-μέλη. Και ήρθα τη μέτωπη με πολύ μεγάλες αντιθέσεις από την Ορθόδοξη Εκκλησία, από την Καθολική Εκκλησία, ιδιαίτερα στην Ανατολική Ευρώπη και δεν ήταν καθόλου εύκολη συζήτηση, αλλά ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για μένα, διότι άκουσα και τις ενστάσεις τους και άρχισα να κατανοώ γιατί υπάρχει τόσος φόβος ε, και ε, υπήρξαν και κάποια επιχειρήματα. Ο διάλογος είναι σημαντικός. Γι' αυτό ακριβώς και στη συνθήκη ε, ο διάλογος με τις εκκλησίες και φιλοσοφικές και μη θρησκευτικέ οργανώσεις προβλέπεται ρητός και σκοπεύω να ε, συμμετέχω. Προβλέπετε δύο φορές το χρόνο. Προσπαθώ να δω με ποιο τρόπο και με ποια μέθοδο θα γίνουν όλα αυτά, αλλά πολύ ευχαριστώ να συμμετέχω σε αυτό το διάλογο. Τώρα, για δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι αυτά είναι θέματα τα οποία δεν είναι στην ε, εντολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γι' αυτό και έχουμε απορρίψει κάποιες τέτοιες πρωτοβουλίες σαν αυτές που αναφέρετε. Θα πρέπει βέβαια να το εξετάσω Θυμάμαι για παράδειγμα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε μια συζήτηση για το νόμο κατά των αμβλώσεων στην Πολωνία. Εγώ ήμουν παρούσα και έπρεπε να πω ότι δεν μπορώ να συμμετέχω ενεργά γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αρμοδιότητα για τέτοιες υποθέσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Σπούρεκ, ένα λεπτό. Εγώ αναφερόμουν σε πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων πολιτών. Αν μπορείτε να μας πείτε λίγα περισσότερα λοιπόν από αυτού. Στις απαντήσεις σας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είπατε ότι εργάζεστε κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού και αυτό για μένα ως πρώην ε, αναπληρώτρια επίτροπο για ανθρώπινα δικαιώματα στην Πολωνία είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πώς σκοπεύετε λοιπόν να αποτρέψετε ξενοφοβικές ε, δυνάμεις ε, να προωθήσουν αντιδημοκρατικά και ρατσιστικά θέματα βάσει και του άρθρου 2 και των αξιών που αναφέρονται στη συνθήκη. Για ένα λεπτό, κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, ε, μια διευκρίνηση. Όποτε λαμβάνουμε μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών και δεν είναι της αρμοδιότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ε, την εξετάζουμε. Αυτό είναι περισσότερο νομικό βέβαια παρά πολιτικό θέμα. Ε, όσον αφορά το ρατσισμό και την ξενοφοβία, είναι πολλά, πάρα πολλά τα πράγματα που κάνουμε. Υπάρχει απόφαση πλαίσιο κατά του ρατσισμού και τη ε, ξενοφοβίας που όπως είπα και προηγουμένως είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα διότι παρακολουθούμε με ποιο τρόπο τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν αυτή την οδηγία και την απόφαση πλαίσιο στην ένωμη τάξη τους. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα για τη στήριξη της κοινωνίας των πολιτών που ε, αφορούν τις μειονότητες και συνεργαζόμαστε και με τις μειονότητες και υπάρχουν και πάρα πολύ σημαντικά προγράμματα που χρωματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να βοηθήσουμε ανθρώπους που βρίσκονται σε κοινωνική ανάγκη και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει για κάποιες μειονότητες. υπάρχουν και εκστρατείε. Εγώ ξεκίνησα προσωπικά την εκστρατεία για την προστασία και την υποστήριξη των ε, ΛΟΑΤΚΙ. Ήταν ε, μια πάρα πολύ χρήσιμη εκστρατεία, πιστεύω, και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Πρέπει να συνεχιστούν όλα αυτά. Και τώρα η συνάδελφος Γκουεντολίν Τελμπό Κάρφιλτ, παρακαλώ. Με ευχαριστώ. Κυρία Γιώροβα, Ακούσαμε από πολλούς ότι το χαρτοφυλάκι όσα θα είναι κομβική σημασίας. Ε, ζούμε δύσκολους καιρούς και κινδυνεύει η δημοκρατία. Για να είναι ζωντανή είναι όλα αλληλένδετα. Ελευθεροτυπία, ε, ελευθερία της έκφρασης, έκφραση των πολιτών, ε, προεκλογικές εκστρατείες, ε, πεντακάθαρες, πολιτική χρηματοδότηση των κομμάτων κτλ. Έγινε μέγας λόγος σήμερα κατά τη διάρκεια της ακρόασης για την παραπληροφόρηση και τους κινδύνους και τους κινδύνους επέμβασης στα προεκλογικά. Συγκεκριμένα, οι ιδιώτες που έχουν πολύ μεγάλα συμφέροντα, όπως είναι κάποιες μεγάλες πολυεθνικές, από όπου και αν προέρχονται, πώς θα μπορούν να αποκλείονται δεδομένης πάντα της ε, ελεύθερης έκφρασης. Οι πλατφόρμες θα πρέπει οι ίδιες να ελέγχουν το περιεχόμενο, να λογοκρίνουν ή να έχουν αλγορίθμους που να μπλοκάρουν το περιεχόμενο αυτόματα. Ή πιστεύετε ότι για, να κλείσουν λογαριασμοί και να καταργηθεί το περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ε, νόμος που παραβιάζεται και να υπάρχει δικαστική απόφαση. Ευχαριστώ ε, κυρία Ντελπός ε, για την ερώτησή σας. Κοιτάξτε να δείτε, ε, πάρα πολύ σύντομα. Εμείς θέλουμε οι πλατφόρμες να συνεργάζονται και να απομακρύνεται το παράνομο ε, περιεχόμενο. Και εδώ μιλούμε για παιδική πορνογραφία, τρομοκρατία, ρητορική μίσους. Αυτοί έχουν τις παραμέτρους ε, για το τι απαγορεύεται από τον ποινικό νόμο σε όλα τα κράτη-μέλη. Και εδώ είμαστε στα χέρια τους. Για τη ρητορική του μίσους που είναι και το πιο λεπτό θέμα, γιατί πολύ σωστά μπορούν να πούν ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Τι θέλουμε να κάνουν οι πλατφόρμες. Να αξιολογούν τις περιπτώσεις και σε περίπτωση αμφιβολίας να είναι υπέρ του ε, λογαριασμού, όπως παραμένει αυτό, όπως στη Γερμανία που έχουν νομοθετήσει. Στη Γερμανία είναι το αντίθετο. Σε περίπτωση αμφιβολίας αφαιρούν το περιεχόμενο γιατί και εμπίπτει στις κυρώσεις. Ε, δεν θέλω να επικρίνω τη Γερμανία, αλλά υπάρχει και η θελοντική δράση υποχρεωτική λόγω του νόμου. Θα δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Θα υπάρξει νομοθεσία που θα προτείνουμε προσεχώς για τις επιγραμμικές υπηρεσίες υπό την αιγίδα της κυρίας Βεστάγκερ και επίσης θα δούμε και τι γίνεται με τους αλγορίθμους. Ε, λειτουργούν. Θέλουμε να έχουμε περισσότερη διαφάνεια εδώ, γιατί θα πρέπει ε, να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος, ε, η ίδια η κατασκευή αυτή και για ποιο λόγο. Γιατί αυτό μπορεί να παραβιάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα και να έχει ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ επιβλαβές προς την κατεύθυνση αυτή. Θέλουμε να μελετήσουμε λοιπόν διάφορα ε, εκεί και πιστεύω ότι η Ευρώπη επιτυχάνει καλά αποτελέσματα. Αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, μια πρόταση ακόμα στα ψηφιακά και στο ε, βλαβερό περιεχόμενο. Η Ευρώπη έχει καλά ένστικτα. Αν το συγκρίνουμε με τις Ηνωμένε Πολιτείε, εμείς θα πάμε πολύ καλύτερα και στην προστασία και στην απομάκρυνση του παράνομου περιεχομένου. Η κυρία Ντελμπός, ε, συμπροματική ερώτηση. Ευχαριστώ για αυτή την πρώτη σας απάντηση. Θα επανέλθουμε σίγουρα και θα σας ξανακάνουμε ερωτήσεις. Ε, κάνατε κάποιες διευκρινήσεις, δεν με καλύπτουν, αλλά θα δείξει. Άλλη ερώτηση τελείως διαφορετική για την Ουγγαρία. Ήδη από την αρχή της ακρόασης ακούσαμε την κατάσταση σε κάποιες χώρες και ιδιαίτερα στην Ουγγαρία. Έχω την τιμή και κυρίως την πολύ μεγάλη ευθύνη να είμαι εισηγήτρια για το Κοινοβούλιο. Η Φιλανδική Προεδρία έδειξε και δείχνει μεγάλη αποφασιστικότητα και δεν ε, ε, μπορούμε παρά να την χαιρετήσουμε. Ε, απαντήσατε στους συναδέλφους Ντόνατ και Ράιντσκε ότι δεν θεωρείται φυσιολογικό το Κοινοβούλιο να μην εμπλέκεται επαρκώς και θυμήσατε πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του στην ενεργοποίηση του άρθρου 7. Αλλά και πάλι δεν σας βρήκα εκεί πολύ αρκετά συγκεκριμένη. Θέλω να ρωτήσω κάτι που ρωτάω πολλούς και άλλοι συνάδελφοι. Θα ήσασταν υπέρ μιας ακρόασης ε, του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. Και όλη αυτή η διαδικασία του άρθρου 7 έχει παραγκονίσει λίγο το Κοινοβούλιο και αυτό μπορεί ε, να φανεί ως απόπειρα ελαχιστοποίησης ε, του ρόλου του. Θα δώσετε τον πλήρη ρόλο που του αναλογεί στο Κοινοβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τους πολίτες. Ευχαριστώ. Είναι η σειρά σα τώρα και πάλι κυρία Γιώργα. Ευχαριστώ πολύ. Θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένω. Στην περίπτωση τη Ουγγαρίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργοποιήσει το άρθρο 7. Βεβαίω συμμετέχει πλήρως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι και λογική όσο και απαραίτητη η πλήρης ε, εμπλοκή του. Και πάρα πολύ σωστή στην ετήσια ε, επισκόπηση του κράτους δικαίου και χάρη ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και χάρη στις συστάσεις που έγιναν We'll try to find θα πρέπει να βρούμε τον καλύτερο τρόπο ε, να σχεδιάσουμε ε, τον τρόπο που θα συμμετέχει το Κοινοβούλιο. Γιατί πραγματικά ε, θέλω να είναι με πλήρη διαφάνεια και να μην γίνονται όλα αυτά κρυπτό και παραβίστο. Πραγματικά είμαι δεσμευμένη προς την κατεύθυνση αυτή, να έχουμε όσο γίνεται ε, πιο στενή και εντατική συνεργασία. Μάλιστα. Η κυρία Μπέρντερ, παρακαλώ, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις περιστατωμένες σας απαντήσεις. Σχεδόν τελειώνουμε. Αλλά ακούσαμε κάποια από τα σχέδιά σας για τη διαφάνεια του νομοθετικού κύκλου. Εγώ θα ήθελα να γνωρίζω πόσο σύντομα σκοπεύετε να ανοίξετε και στον έλεγχο τους τριμερίους διαλόγους, γιατί όπως ξέρετε ε, πολύ μας ενδιαφέρει η διαφάνεια εδώ, καθώς αναπτύσσουμε και τη σχετική νομοθεσία. Ε, επίσης έχετε αναλάβει την καλύτερη νομοθετική διαδικασία αλλά όσο καλή και αν είναι η νόμη, ε, δεν έχουν νόημα και χάνουν την αξιοπιστία ενώπιον των πολιτών όταν αυτοί οι νόμοι ε, παραβλέπονται ή παραβιάζονται και επιβάλλονται ισνά πρόστιμα. Αυτό σημαίνει ότι ε, αποδυναμώνονται οι αξίες που μας είναι εμάς προσφυλής. Η καλή νομοθεσία συμβαδίζει με την επιβολή του νόμου. Τι βήματα θα κάνετε ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η επιβολή του νόμου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σκοπεύετε σκοπεύετε να δημοσιεύσετε την πρόοδο σας σε αυτό το τομέα στην ετήσια έκθεση περί επιβολής της νομοθεσίας. Κυρία Γιούροβα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μπίρντερ για τις ερωτήσεις σας. Καταρχάς διαφάνεια. Θα ήθελα να... Υποβάλλω αρχικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσα στο χρόνο θα πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Είναι ένα από τα ε, καθήκοντα κλειδιά για μένα, οπότε θα πρέπει αμέσως να αρχίσω να εργάζομαι από αυτών των ζητημάτων. Ίσως να έχουμε κάποια μερικά αποτελέσματα το επόμενο εξάμεινο. Ε, δεν βλέπω λόγο δηλαδή να καθυστερούμε ούτε να περιμένουμε γιατί η διαδικασία αυτή είναι διαρκής, είναι συνεχής. Μιλώντας για διαφάνεια και διαφανή νομοθετική διαδικασία, δεν χρειαζόμαστε τώρα, χρειάζεται τώρα να βελτιωθεί. Οπότε εκεί θα ενεργήσουμε γρήγορα. Για την καλύτερη νομοθετική δικασία. Ξέρετε ότι έχουμε αυτή την αρχή μια νομοθεσία, εισάγεται μία πάβη. Ε, ε, θα πρέπει όμως να δούμε ποιες είναι οι οδηγίες οι οποίες ε, δεν πληρούν πια το σκοπό για τον οποίο αρχικά ε, συντάχθηκαν. Πρέπει να είμαστε θαραλέοι. Πρέπει να ξεφορτωθούμε όλες εκείνες τις νομοθεσίες από τη δεκαετία του 80 που δημιουργούν μεγάλο φόρτο για τις μικρομεσαίες. Θα πρέπει δηλαδή να ε, κάνουμε περισσότερα και ναι, μπορεί όλα αυτά να δημοσιευθούν στην ετήσια έκθεση πρόοδου. Κυρία Μπέρντερ, έχετε ένα δεύτερο λεπτό. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας, αλλά όσον αφορά την επιβολή δεν τα πάμε καλά. Να αναφέρω μόνο τη Volkswagen, τη συνεχιζόμενη... Ε, ε, ε, θανάτωση των μεταναστευτικών, των αποδημητικών πουλιών, ένα σωρό όλα πράγματα. Και οι πολίτες παρακολουθούν, φτιάχνουμε νομοθεσίες και μετά τα κράτη-μέλη συνεχίζουν ε, το χαβά τους. Ε, βεβαίως ε, θα πρέπει να καταλάβετε ότι εμείς ε, προσβλέπουμε σε εσά και σε εσά δηλαδή κυρία υποψήφια να σταθείτε, να ορθώσετε το ανάστημα της Ένωσης όταν παραβιάζετε την νομοθεσία. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι είστε προσιλωμένοι στην επιβολή του νόμου στα κρατημέλη. Ναι βεβαίως. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει να είμαστε όσο γίνεται πιο διαφανείς σε αυτά τα θέματα. Τουλάχιστον εγώ αυτό έκανα στο δικό μου το ε, ε, χαρτοφυλάκιο. Ποτέ δεν ε, δίστασα να δακτυλοδείξω τα κράτη-μέλη που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Θα το κάνω και στο μέλλον. Θα είναι πρακτική μου και θα είμαι εκείνη που θα πιέζει για όσο το δυνατόν περισσότερη διαφάνεια στην εφαρμογή του νόμου. Μάλιστα. Και τώρα για να ολοκληρώσουμε το γύρο των 25 ερωτήσεων, Τελευταίο ομιλητή μα θα είναι ο συνάδελφος Λοράν. Ευχαριστώ. Ω τελευταίο δύσκολο μπορώ να προσθέσω κάτι, αλλά θα προσπαθήσω. Ο κύριο Βίντσε. Κυρία Γιούροβα, είστε υπεύθυνη για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών ισχύει εδώ και 7 χρόνια και δεν έχουν ε, και πολλά αποτελέσματα. Από τις 70 προτάσεις μόνο 6 ε, ξεκίνησαν. Θα υπάρξει νέα νομοθεσία ώστε να είναι πιο εύκολα και πιο απλή η διαδικασία για τους πολίτες. Η εμπειρία δείχνει, όπως είπατε και εσείς σήμερα, ότι οι βασικές προκλήσεις για τη διαδικασία των πολιτών δεν είναι μόνο η διαδικασία και οι ε, απαιτήσει, αλλά η διστακτικότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προωθήσει τις ε, προτάσεις αυτές. Ε, μέχρι τώρα καμία από τις τέσσερις νομοθετικές προτάσεις ε, δεν έγινε νομοθετική πράξη. Υπάρχει δηλαδή ένα δικαίωμα για τους πολίτες από τη συνθήκη της Λισαβόνας που δεν έχει εφαρμόσει ούτε μία φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τι θα κάνετε λοιπόν προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι οι πρωτοβουλίες των πολιτών δεν θα είναι απλώς μία συμβολική πράξη συμμετοχή στη δημοκρατία. Έχετε το λόγο κυρία Γιούροβα για να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βίντσε για την ερώτησή σας. Χαίρομαι που το ρωτάτε αυτό, διότι όταν είδα στην επιστολή των καθηκόντων μου ότι έχω και την πρωτοβουλία των πολιτών, αμέσως άρχισα να σκέφτομαι πώς θα μπορέσω να μετατρέψει αυτή την τυπική διαδικασία σε κάτι ζωντανό, κάτι πιο πρακτικό για τους πολίτες ε, ε, και κάτι που θα είναι πολλά υποσχόμενος προς την επικοινωνία. Είναι πολύ σωστά τα στοιχεία σας, δεν ε, ελήφθησαν πολλές υπόψεις για συνέχεια. Δεν συμφωνώ όμως ότι δίστασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεχτεί τις προτάσεις. Θα έλεγα μάλλον ότι η διαδικασία ήταν αρκετά χρονοβόρα και νομικίστικη και αφορά και τη επικοινωνία με τους διοργανωτές ε, αυτό. Θα ήθελα να το αλλάξω. Θα κάνω χρήση της νέας νομοθετικής εκδοχής ε, της ε, πρωτοβουλίας των πολιτών, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από πρώτης πρώτου. Πρέπει να επιταχύνουμε την επικοινωνία, πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα το ηλεκτρονικό σύστημα για την επικοινωνία με τους διοργανωτές και θα εξετάσουμε και το ενδεχόμενο να υπάρχουν κάποιες γραμμές βοήθειας ε, και κάποια υποστήριξη, ώστε αυτοί οι οποίοι θέλουν να υποβάλουν μια πρωτοβουλία πολιτών να ξέρουν τι να κάνουν όσον αφορά τις τυπικές υποχρεώσεις. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να αντιστρέψω την κατάσταση. Ευχαριστώ. Τελευταία συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Βίντσε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας, κύριε Επίτροπε για να συμπληρώσω την ερώτησή μου μάλλον μια προηγούμενη ερώτηση. Αυτή τη στιγμή σε κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν νόμοι για την προστασία εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων, αλλά δεν εφαρμόζονται όλοι ή εφαρμόζονται μερικώς. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός κράτους δικαίου και παρακολούθησης που θα εξετάσει και την παρούσα νομοθεσία για τον τομέα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων πιο συγκεκριμένα. Έχετε το λόγο κυρία Γιούροβα. η αξιολόγηση και οι πιθανές ε, δράσεις ε, κατά την άποψή εντάσσονται περισσότερο στην, ε, στο θεματολόγιο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και όπως σα είπα, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για την εφαρμογή του χάρτη. Θα εξετάσουμε πώς εφαρμόζεται και αυτό σημαίνει ότι θα εξετάσουμε και τον τρόπο με τον οποίο προωθούμε τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και πώς εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία σε επίπεδο κρατών μελών. Πιστεύω ότι ε, θα είναι πιο ισχυρή η εξέταση μέσω των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπου θα δούμε τα δικαιώματα των μειονοτήτων και τις γλωσσικές μειονότητες. Πολύ σημαντικός γύρος, 25 ερωτήσεις, ε, ετέθησαν όλες, απαντήθηκαν όλες. Φτάνουμε λοιπόν στο τελευταίο σκέλος της ακρόασης, που περιλαμβάνει να δώσουμε και το λόγο στην ε, υποψήφια αντιπρόεδρο ε, της Επιτροπής, την κυρία Γιούροβα. Έχετε το λόγο για να κάνετε την τελευταία σας παρέμβαση πριν ολοκληρωθεί η ακρόαση και πριν ε, εγώ και ο συμπρόεδρος, ο κύριος Σταγιάννη, ανακοινώσουμε τι θα γίνει στη συνέχεια για τη συνεδρίαση των συντονιστών για την αξιολόγηση. Παρακαλώ. Αξιότιμη πρόεδροι, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση αυτή. Πιστεύω ότι ήδη από τώρα μπορώ να πω έτσι ενθερμώ ότι δύο πράγματα με επιβεβαίωσε η παρούσα ακρόαση. Πρώτον, ότι όλες οι επιτροπές ε, έχουν πολύ αξιόλογα μέλη που θα εργαστούν σκληρά την επόμενη πενταετία για όλα αυτά τα προβλήματα και τα θέματα. Και είναι πάρα πολύ καλό που αισθάνομαι ότι έχω ισχυρούς συμμάχους εδώ στο Κοινοβούλιο. Το δεύτερον, η εκλεγμένη πρόεδρος Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν από την αρχή θέλησε να δημιουργήσει ένα χαρτοφυλάκιο με τη δική μου περιγραφή των καθηκόντων. Είναι νέο αυτό το χαρτοφυλάκιο, δεν υπήρχε στο παρελθόν και ε, βγάζει συμπεράσματα από τις νέες προκλήσεις που έχουμε, τις νέες απειλές για τη δημοκρατία μας. Οι παλιές απειλές διευρύνονται με νέα μέσα και τις νέες τεχνολογίες. Επίσης βλέπουμε ε, προκλήσεις, στις ε, ίδια τα θεμέλια στα οποία ε, έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τα θεμελιώδη δικαιώματα βλέπουμε ότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος λήψης αποφάσεων για να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και να κατανοούν καλύτερα και πιο εύκολα οι πολίτες όλα αυτά. Θα πρέπει να εξοπλιστούμε εν ώψη των εκλογών του 2024, γιατί διακυβεύονται πολλά και εάν μας νοιάζει θα πρέπει να τολμούμε. Δεν είναι το τέλος της ιστορίας, σε αντίθεση με όσα είπε ο Φουκουγιάμα. Ίσα ίσα ε, ε, η ιστορία όχι απλώς ε, δεν έχει τελειώσει, αλλά επιταχύνεται κιόλας. Ρόλος μου θα είναι να συντονίσω το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να είμαι ο μεγενθητικός φακός για οτιδήποτε κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να επαγρυπνώ για το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ότι θα πρέπει να είναι από το σχεδιασμό σε όλους τους τομείς πολιτικής και η δημοκρατία μας να αυξάνεται και να γίνεται όλο και πιο ανθεκτική απέναντι στις σύγχρονες απειλές. Επίσης θα εργαστώ πολύ στενά, θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους, ιδιαίτερα με τον Επίτροπο Αρμόδιο για τη Δικαιοσύνη και θα χρησιμοποιήσω αυτό τον οριζόντιο ρόλο μου για να σπάσω τα στεγανά και να φέρω κάτω από την ίδια στέγη όλες τις πολιτικές. Μου εμπιστεύτηκε να δώσω ζωή σε νέες ιδέες η κυρία Φόντερ Λάιν, όπως ε, ε, ο νέος μηχανισμός για το κράτος δικαίου ή το πρόγραμμα δράσης για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Είμαι ισχυρό, συνήγορος των πολιτών. Έτσι αντιλαμβάνομαι το ρόλο μου. Θέλω να ακούγονται οι πολίτες ατομικά και συλλογικά και να μην αγνοείται η φωνή τους και θα πρέπει τα δικαιώματά τους να γίνονται σεβαστά και όχι να καταπατώνται. Θέλω να αγωνιστώ ε, ώστε οι πολίτες να εμπιστεύονται την Ευρώπη, βελτιώνοντας τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε τους ηγέτες μας και να έχουμε για όλες τις ε, θέσεις ε, ισχυρά κριτήρια. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ένα πράγμα είναι για μένα ξεκάθαρο. Δεν θα μπορέσω όλα αυτά να τα κάνω μόνη μου. Όλα τα βήματα μας ε, απαιτούν δημιουργικότητα, διακομματική συνεργασία και αποφασιστικότητα. Ε, είμαι προσιλωμένη στη συνεργασία μας και μπορώ σίγουρα να προσβλέπω στην υποστήριξή σας, στο αυστηρό σας μάτι και στις ιδέες σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία υποψήφια την Πρόεδρε Γιούροβα. Ευχαριστούμε και όλα τα μέλη που συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε όλες για την προετοιμασία και για τις ερωτήσεις που ακούσαμε μέχρι τώρα. Φτάνουμε στο τέλος τώρα και είναι η στιγμή να πούμε τα τελευταία πράγματα. Θα είδατε ότι το όνομα του χαρτοφυλακίου σα αποτελεί πρόκληση για όλες μας, αξίες και διαφάνεια, γιατί και τα δύο είναι χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής διαδικασίας του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Ακριβώς όμως γι' αυτό το λόγο ε, υπόκειται και σε νέε προκλήσεις οι οποίες ε, δημιουργούν και νέε απειλέ που σημαίνει ότι χρειαζόμαστε νέε ικανότητες. Η ψηφιακή εποχή που είναι και το όνομα ενό σημαντικού χαρτοφυλακίου άλλου αντιπροέδρου αυτή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα δημιουργήσει νέε προκλήσει για τον τρόπο με τον οποίο έχουμε βιώσει τη δημοκρατία και την πολιτική συμμετοχή και την ηθαγένεια μέχρι τώρα. Όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης που αδιαμφισβήτητα είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη, αυτό ενισχύεται από την ψηφιακή εποχή, αλλά και ε, είναι και έρμεο νέων απειλών και προκλήσεων, γιατί μπορεί να υπάρξει χειραγώγηση και παραπληροφόρηση από τα μέσα ε, κοινωνική δικτύωση που μπορεί να δημιουργήσει και στρέβλωση τη δημοκρατικής ε, διαδικασίας ε, και τη διαδικασία του νόμου και της ίδιας ουσίας του κράτους δικαίου. Είναι πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση λοιπόν, διότι θα πρέπει να συντονίσετε και άλλε σημαντικέ πτυχές της μελλοντική Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μα έχετε αποδείξει ότι ενδιαφέρεστε, σα γνωρίζουμε, έχουμε μάθει να γνωρίζουμε πράγματα για εσά, γιατί πολλοί από εμά που ανανέωσαν τη φοιτεία τους εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας γνώρισαν την προηγούμενη πενταετία, σας έχουμε δει και επί το έργο και σίγουρα θα επαγρυπνούμε για το τι μελιγενέστε, διότι το μόνο προφανές είναι ότι η νέα δομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα δημιουργήσει προκλήσεις όχι μόνο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πώς θα ε, συντονίζεστε και θα συνεργάζεστε μεταξύ σας Υπάρχουν τομείς ε, που έχουν επικαλύψεις και θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο συντονισμός ε, με τα διάφορα χαρτοφυλάκια και με τους υπόλοιπους ε, επιτρόπους, ώστε όλη η δουλειά πραγματικά να έχει και κάποιο νόημα. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε για την προσπάθειά σας και την ενέργεια που αφιερώσατε εδώ τις προηγούμενες δυόμιση ώρες και τώρα να δώσω το λόγο στον συμπρόεδρό μας, τον πρόεδρο Ταγιάννη, από την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων, ώστε να ολοκληρώσω και τη συνεδρίαση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπες Αγγελάρα. Να καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές που προέρχονται από τις Επιτροπές ΑΦΚΟ, ΛΥΜΠΕ και Τζούρι. Να ευχαριστήσω τους διερμηνείς. Χάρη σε εσάς μπορούμε να μιλάμε όλη αυτή την ώρα. Επίσης ε, και αυτό υπερασπίζει τη δημοκρατία, όπως είπε και ο συνάδελφος ε, Αγγιλάρα, ε, πρέπει να στηρίξουμε την ελευθεροτυπία. θυμίζουμε πως η Αλήσια η Καρουάνα Γαλήσια δολοφονήθηκε. Δολοφονήθηκαν δύο δημοσιογράφοι στο Στρασβούργο πέρσι τα Χριστούγεννα. Ε, πρέπει αυτό να το κάνουμε Όχι αυτό δεν το λέω επειδή είμαι δημοσιογράφο, αλλά επειδή πιστεύω πω η ελευθεροτυπία είναι θέμα κλειδί για τη δημοκρατία και για τη διαφάνεια χρειάζεται, χρειάζεται η δέσμευσή μας όχι μόνο ε, με τα λόγια αλλά με τις πράξεις ε, Τέλος Η συνεδρίαση ανάμεσα στους συντονιστές της ΑΦΚΟ και της ΛΥΜΠΕ θα λάβει χώρα στις 6 και 30 μετά από μια σύντομη συνέντευξη τύπου, δήλωση τύπου 6 και 30 το βορρά το απόγευμα. Είμαστε έτοιμοι και αύριο το πρωί συνομιλία εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους. Πέρα στη συζήτηση. Okay.